Good morning. Καλή σας μέρα. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης και θα μιλάω ισπανικά. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Τώρα θα εξετάσουμε το κείμενο για την Τουρκία, την 2015 για την Τουρκία. συνολική στρατηγική. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πύρη. Με τους εναλλακτικούς, ε, συγγνώμη, τους ε, εξέτασαν ε, τις τροπολογίες. Υπάρχουν 37 συμβαστικές που αναφέρονται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και συμπεριλαμβάνεται και συνεργασία στα θέματα μετανάστευσης, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Επιπλέον, αναφέρεται και η ενισχυτική κατάσταση στην υπόλοιπη Τουρκία και οι συζητήσεις όσον αφορά την ενοποίηση της Κύπρου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Πύρη για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πριν αρχίσουμε τη δεύτερη εξέταση της έκθεσης του 2015 για την Τουρκία, επιτρέψτε μου να εκφράσω εδώ τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στα, στις οικογένειες των θυμάτων της τελευταίας τρομοκρατικής επίθεσης στην Άγκυρα. Και μιλάω εκ μέρους όλων μας όταν λέμε ότι πενθούμε μαζί με τον τουρκικό λαό και επαναλαμβάνουμε την ε, πεποίθησή μας ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Πρόεδρε, συνοψίσατε πολύ καλά τα πράγματα. Σήμερα με τους ε, σκιώδες συζητητές από τις άλλες πολιτικές ε, ομάδες συζητάμε το θέμα αυτό. Έχουμε 37 συμβιβαστικές τροπολογίες, τις τελευταίες εβδομάδες καταλήξαμε σε αυτές και θέλω να εκφράσω την ευγνώμοσύνη μου σε όλους τους γιατί τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή που μπορεί να υποστηριχθεί τελικά από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κύρια συμπεράσματα στην ε, έκθεση που θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα στην Επιτροπή μας περιλαμβάνονται στις 37 συμβαστικές τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια γενική σοβαρή ανησυχία όσον αφορά το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων που επιβραδύνθηκε γενικά και σε ορισμένους τομείς όπως είναι η ελευθερία έκφρασης ή η ανεξαρτησία τους δικαιοσύνης έχουν πάει πίσω αντί να πηγαίνουν μπροστά. Υπάρχει τεράστια πίεση από την κυβέρνηση σε κάθε έκφραση κριτικής, είτε προέρχεται από δημοσιογράφους, όπως το είδαμε με το κλείσιμο της εφημερίδας ε, Ζάμων και της Υπηρεσίας Νέων, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις το διαπιστώνουμε αυτό. Ακαδημαϊκοί που μιλούν υπέρ της ειρήνης, ε, υπάρχει εκφοβισμός και σε βάρος των μελών της αντιπολίτευσης, σε καθημερινή βασικά βάση. Από εκεί ξεκινάει η έκθεση λοιπόν. Έπειτα κάνει έκκληση να σταματήσει η βία στα Ανατολικά και να αρχίσει και πάλι ο διάλογος. Καταδικάζουμε την επιστροφή της βίας από το ΠΚΚ που βρίσκεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η, η κατάπαυση πυρός που έχει αποφασιστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και το κράτος τελικά ο κόσμος που ζει στις ε, κουρδικές ε, αυτές περιοχές, 350.000 σύμφωνα με το ίδιο το κουρδικό Υπουργείο, πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους, κάτι το οποίο βέβαια οδηγεί σε μεγάλη ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία. Και κάνουμε και έκκληση για να εντατικοποιηθεί ο διάλογος για όλα αυτά τα ζητήματα και ο καλύτερος τρόπος είναι ο διάλογος αυτός να λάβει χώρα στα πλαίσια της διαδικασίας ε, ένταξης. Βέβαια εδώ έρχομαι και σε αυτό που θα συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή για την μετανάστευση. Εμείς ε, λέμε μπράβο στη, στον τουρκικό λαό για το βάρος που έχει αναλάβει που είναι το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων. Όντως πρέπει να βρίσκουμε λύσεις στην προσφυγική κρίση. Αλλά εδώ οι διάφορε πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν οι προσπάθειε αυτέ να συνδυαστούν, μάλλον να μην συνδυάζονται, να μην συνδέονται με τις συνομιλίες που έχουμε για ένταξη της Τουρκίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι κάτι που μπορείτε να διαπραγματευτείτε όταν μιλάτε για την μετανάστευση στο προσφυγικό. Και εδώ ο διάλογος με την τουρκική κυβέρνηση δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσοι φτάνουν στα ελληνικά νησιά κάθε μέρα από την Τουρκία. Πρέπει να δούμε και τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία οι προδιαγραφές ας πούμε όσον αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης θεωρήσεων είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη και ζητάμε από την ε, τουρκική κυβέρνηση να λάβει υπόψη στη σύμβαση της Γενέβης οπότε να μπορούν να ζητήσουν ε, και Ιρακινοί και Αφγανοί άσυλο. Επίσης χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επανένωση της Κύπρου. Υπογραμμίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που κρατάει εδώ και δεκαετίες και που είναι πολύ σημαντικό για όλη την περιοχή και βέβαια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από την Τουρκία και όλους τους διεθνείς εταίρους να προσεγγίσουν θετικά τη διαδικασία αυτή και τέλος για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας και το προσωπικό όλων των πολιτικών ομάδων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων επειδή σε βάση 24 ώρου, με full time μας υποστήριξαν, μας βοήθησαν για να μπορέσουμε να έχουμε σήμερα το πρωί αυτή τη συζήτηση και το απόγευμα την ψηφοφορία. Αυτά είχα να πω πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Πύρη. Θα δώσουμε το λόγο τρία λεπτά στο κάθε σκιώδη Ο κύριος Σόμερ είναι ο πρώτος από το Η κυρία Σόμερ, διορθώνει ο πρόεδρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους ε, συγγενείς ε, των ε, θυμάτων της τελευταίας κομμουνιστικής επίθεσης στην Τουρκία και ελπίζω ότι θα καταφέρει η Τουρκία να μην συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, αλλά βέβαια ζούμε σε μια πολύ ανασφαλή και βέβαια περίοδο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την συγκεντρία κυρία Κατυπήρη, αλλά και τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ε, ήταν ε, πραγματικά ασφικτικά τα χρονικά μας περιθώρια. Είχε αρχικά προβλεφθεί μόνο μία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να βρούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς, αλλά είναι τόσο περίπλοκο το ζήτημα και ήταν τόσο υψηλός ο αριθμός, περίπου 550 τροπολογίες κατατέθηκαν. Ήταν τόσο λοιπόν ο αριθμός που δεν ε, περιοριστήκαμε μόνο σε μία συνάντηση, αλλά κάναμε τρεις συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και συμφωνήσαμε επί της αρχής να ακολουθήσουμε τη γραμμή, αν θέλετε, που είχαμε ακολουθήσει και πέρυσι. Και ίσως η διαπραγμάτευση ε, μας διευκόλυνε ακριβώς το να τηρήσουμε την ίδια αυτή γραμμή. Πράγματι η κατάσταση στην Τουρκία δεν έχει μεταβληθεί, δεν διακρίνουμε κάποια δηλαδή πρόοδο, πρόοδο σε ό,τι αφορά την, τον εξευρωπαϊσμό αν θέλετε της Τουρκίας. Αντιθέτως ε, βλέπουμε να υπάρχει μια επαναχώρηση, οπισθοδρόμηση αν θέλετε, που παρατηρείται και από, στην έκθεση της Επιτροπής ε, και βέβαια είναι ε, ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι την προηγούμενη μέρα πριν από τη σύνοδο της κορυφής η Ζαμάν ε, τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο και την ημέρα της Συνόδου Κορυφής ένας ακόμα φορέας τέθηκε υπό τον κρατικό έλεγχο. Αυτά λοιπόν ε, μας δείχνουν ότι η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει από την πλευρά της δηλαδή. Ό,τι και αν εμείς κάνουμε η Τουρκία παραμένει η ίδια, ακολουθεί την ίδια πολιτική και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σκέφτεται τουλάχιστον η Τουρκία, θα πρέπει να τα αποδεχτεί όλα αυτά γιατί εξαρτάται από την Τουρκία, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική κρίση. Όμως εμείς ε, θεωρούμε όλοι από την πλευρά δηλαδή των ΣΕΙΤΟΝ, ε, ότι δεν θα πρέπει ακριβώ να αναμειγνύουμε αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή τη μεταναστευτική κρίση αφενό και τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει τη Τουρκία. Δηλαδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εκπτώσει εντό εισαγωγικών ε, στην Τουρκία για να επιλύσουμε τη μεταναστευτική κρίση. Φυσικά θέλουμε μια καλή συνεργασία με την Τουρκία, αλλά δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να μα ασκήσει πιέσει και νομίζω πω αποτελεί καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το καταδείξει αυτό. Ότι δηλαδή ναι, βρισκόμαστε υπό πίεση ακριβώ λόγω του μεταναστευτικού τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωση και η ίδια Ένωση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τέτοιου είδου παραχωρήσει και ε, ε υιοθετώντα ένα σχετικό ψηφίσμα. Ε, βέβαια τώρα στην ε, έκθεση υπήρχαν κάποια αρκετά περίπλοκα ζητήματα, ειδικότερα το ζήτημα τη Κύπρου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και έχει προτεραιότητα και αποτελεί βέβαια και ε, αν θέλετε το, ένα ιδιαίτερο τεστ για το, πώς, ε, για το σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένη και ικανή να επιλύει τα προβλήματά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να προδικάσουμε την λύση η οποία θα επιτευχθεί σε σχέση με το Κυπριακό. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε ένα separate constituent state όπως αναφέρεται μέσα σε αυτό το κείμενο. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητο να γίνεται μια τέτοια αναφορά ή για παράδειγμα ε, το, να συμπεριλαμβάνεται ως επίσημη ή όχι γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα τουρκικά. Δεν νομίζω ε, πως χρειάζεται να γίνεται μια τέτοια αναφορά. Δηλαδή με, κάτι, με μια τέτοια αναφορά ουσιαστικά προδικάζουμε το αποτέλεσμα μια συζήτηση η οποία ακόμα βρίσκεται μπροστά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη γραμματεία της Επιτροπής μας γιατί ξέρω ότι βρέθηκε υποψηλή ε, πίεση χρόνου και βλέπω ότι και εγώ βέβαια θα πρέπει να ολοκληρώσω. Μου κάνει συνέχεια νόημα ο πρόεδρο ότι θα πρέπει να ολοκληρώσω. Κλείνω λοιπόν εδώ και ελπίζω ότι πραγματικά θα φτάσουμε ένα καλό αποτέλεσμα μετά από τι διαπραγματεύσει μα. Ευχαριστούμε κυρία Σόμερ. Έχουμε πολλού στο κατάλογο μιλητών. Θα κλείσω τώρα το κατάλογο μιλητών και παρακαλώ του συναδέρφου να τηρούν το χρόνο του. Ο κύριο Λάγκστορφ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να εκφράσω καταρχήν τα συλληπιτήρια της ε, πολιτικής μου ομάδας για τα ε, θύματα και τους εγγενείς των θυμάτων ε, στις επίθεσεις στην Άγκυρα που είναι βέβαια τρίτη επίθεση. Πραγματικά η κατάσταση στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί πολύ για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν απλά να ζήσουν καθημερινά τη ζωή τους, δηλαδή διέπεται από φόβο πλέον. Και αυτό αφορά βέβαια την Τουρκία αλλά ειδικότερα και τις πολιτικές ε, περιοχές. Τώρα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ίδιο τη ε, έκθεση. Να ευχαριστήσω λοιπόν την συνάδελφο Ζόμερ, την προφανώ την ε, Κατυπήρ και του υπόλοιπου ε, στιώδει εισηγητέ και την συνάδελφο η οποία με εκπροσώπησε σε κάποιε από τι συναντήσει των στιωδών εισηγητών. Νομίζω πω καταφέραμε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά τρία σημεία θα ήθελα να θέσω που είναι σημαντικά για μα. Στην τροπολογία 9 αναφέρεται ότι θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η διαδικασία τη προσχώρηση και νομίζω πω αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, αν πραγματικά η λόγω διαδικασία αυτή ε, της ε, ενταξιακής διαπραγμάτευσης αποτελεί ε, ένα εργαλείο το οποίο έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί αυτή την περίοδο για τη συνεργασία μας με την Τουρκία. Ένα δεύτερο σημείο. Η συμβαστική τροπολογία 17 και η αναφορά εκεί που γίνεται ε, της ε, βίαιης ε, και παράνομης θέσης υπό κρατικό έλεγχο των εφημερίδων όπως Ζαβάν είναι ενδεδειγμένη. Δηλαδή θα πρέπει να υποθεί με αυτόν τον κατηγορηματικό τρόπο. Η ελευθερία δηλαδή του, του τύπου και ελευθερία της έκφρασης τόσο online όσο και offline αποτελούν πραγματικά ορόσημα των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε τώρα πως υπάρχει μια υποψήφια προσένταξη χώρα η οποία ε, το λόγο και περισσότερο από αυτές τις αρχές. Ένα τρίτο τώρα το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι η ε, συμβαστική τροπολογία 31. Νομίζω πως ε, εδώ συμφώνησαν όλες οι πολιτικές ομάδες ότι δηλαδή το ζήτημα της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμεινέται με την ενταξιακή διαδικασία. Η μεταναστευτική κρίση προφανώς μας θέτει προκλήσεις σε πολιτικό επίπεδο και προφανώς εγώ δεν έχω ε, καμία αντίρρηση απέναντι σε μια εταιρική σχέση με την Τουρκία αλλά όχι με αντίτυπο ε, το να ε, ουσιαστικά να μην τηρήσει, να μην συνεχίσει να τηρεί τις αρχές που έχει θέσει τον εαυτό της Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα σε σχέση και με τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Κάτι ε, τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με έκθεση προόδου, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με έκθεση οπισθοδρόμησης και όπως είπε και η κυρία δεν αντιλαμβανόμαστε κι εμεί γιατί μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λήφθη ένα, ένα τόσο δραστικό μέτρο. Μετά σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτο των ε, θεωρήσεων είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί. Δηλαδή, ανάλογα με τη συνεργασία μα με την Τουρκία θα πρέπει να κινηθεί και η διαδικασία τη ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά σίγουρα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επιτύχουμε πρόοδο γιατί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτε να ταξιδεύουν χωρί προβλήματα και έχουμε και κάποιους εκπροσώπους εδώ της του Ιδρύματος Ευνερμών που είναι ε, ένας φορέας ε, της ε, Τουρκίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Τάξη έχει τώρα το λόγο. Επειδή η επανάληψη των συλληπιτηρίων προς την Τουρκία μπορεί να δώσει προς τους Τούρκους πολίτες και τους συγγενείς των θυμάτων μπορεί να δώσει την εντύπωση μιας διαδικαστικής προσέγγισης του ζητήματος Θέλω να πω και από μέρους μας ότι τα συλληπιτήρια είναι ειλικρινή κυρίως προς τους συγγενείς των θυμάτων. Εγώ από την πρώτη στιγμή έστειλα συλληπιτήριο μήνυμα στον πρέσβη της Τουρκίας στις Βρυξέλλες εκ μέρους εμού και του κόμματος μου βέβαια για αυτή την τραγική εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέχεια προηγούμενων βομβιστικών επιθέσεων. Δυστυχώς αυτές οι βομβιστικές επιθέσεις επιτείνουν το κλίμα ανησυχίας που μας συνέχει ένα και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα η οποία κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ε, χωρίς καμιά αμφιβολία εκτείνεται ε, στα σύνορα της χώρας με πολύ μεγάλα προβλήματα και και της μεγάλης ροής ε, προσφύγων προς την Ευρώπη. Η, η πόλη της Σούρ, την οποία επισκεφτήκαμε πρόσφατα μια αντιπροσωπεία βουλευτών και από ό,τι έχω ενημερωθεί μια νέα επίσημη αποστολή θα επισκεφτεί την περιοχή, βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και 100 μέρες και όπω έχει πει και η συνάδελφο η συγγήτρια τη Έκθεση, η κυρία Πύρη, έχουμε ήδη 350.000 περίπου ανθρώπου οι οποίοι έχουν φύγει από τα σπίτια του. Αυτή είναι μια κατάσταση για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει γρήγορε αποφάσει πίεση προ την κατεύθυνση τη Τουρκία να αρχίσει συνομιλίε ε, για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δυστυχώς θα έχουμε και άλλες, το απέφχομαι, βομβιστικές επιθέσεις και νέους πρόσφυγες που πιθανόν να τους δούμε να παίρνουν τα πόδια τους να έρχονται και αυτοί προς την Ευρώπη. <clears throat> Το κλείσιμο της εφημερίδας Ζαμάν και η καταπίεση, για να μην πω η απαγόρευση κάθε ελεύθερης φωνής στην Τουρκία είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδείξει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό και το οποίο βεβαίω εμπεριέχεται στην έκθεση. Η δίωξη των ακαδημαϊκών, αγαπητοί φίλοι. Χίλια ακαδημαϊκοί υπέγραψαν ένα έγγραφο που ζητά ε, συνομιλίες ειρηνευτικές στο θέμα της, ε, του κουρδικού ζητήματος και όλοι αυτοί οι άνθρωποι διώκονται. Πολλοί εξ αυτών έχουν χάσει ήδη τις δουλειές τους. Θέλω να συγχαρώ σε αυτό το σημείο την Κατυπήρη διότι ε, κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια και ειλικρινή προσπάθεια για δίκαιες συμβιβαστικές ε, σκέψεις ε, προς την κατεύθυνση της υιοθέτηση της, της έκθεσης, αν είναι δυνατόν, με ένα συλλογικό τρόπο. Εμείς δεν έχουμε τίποτα ενάντια στον τουρκικό λαό, όπως δεν έχουμε τίποτα ενάντια σε οποιονδήποτε λαό. Αντίθετα, αγωνιούμε μαζί με τον τουρκικό λαό για το γεγονός ότι υπάρχει πλέον στην τουρκική πρωτεύουσα ένα εργοστάσιο που παράγει φόβο. Τον εγκυτιώνει και τον παραδίδει στα σπίτια των πολιτών. Και όταν συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι ψηφίζουν το κατεστημένο. Θέλω να πω ότι όσον αφορά την Κύπρο, οι αναφορέ είναι ε, σχεδόν στο σύνολό του προ σωστή κατεύθυνση και τη στηρίζομαι απόλυτα. Έχουμε μια έγνοια και αναμένουμε το απόγευμα να υπερψηφιστεί η τροπολογία που αναφέρεται στου έπικου και στην άλλη τροπολογία που αναφέρεται ότι η λύση πρέπει να συνάδει με τι βασικέ αρχέ και αξίε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω με το εξή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω εκεί θα καταψηφίσουν την αναφορά για μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία την ώρα που είναι οι υπερασπιστές της άποψης ότι τέτοια λύση, τέτοια μετεξέλιξη δεν θα υπάρξει με τη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βαλέρο, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς οικογένειες των θυμάτων στην τελευταία αυτή επίθεση στην Άγκυρα. Θα ήθελα όμως παράλληλα να εκφράσω τα βαθύτερά μου αισθήματα για όλους τους ανθρώπους που πρέπει καθημερινά να βιώνουν την κατάσταση αυτή. Και αυτό πρέπει να αναφέρουμε στον πόλεμο αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ερντογάν και Κούρδων. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους. Τίθενται επίσης και κάποιες σημαντικές προτεραιότητες λόγω της επικαιρότητα. Πρέπει πάντως να καταφέρουμε να σταματήσουμε όλες αυτές τις πράξεις βίας, οι οποίες λαμβάνουν πλέον καθημερινά χώρα στην Τουρκία και θέτουν την όλη χώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό στην έκθεση αυτή να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε σε κάποιες βασικές προειδοποιήσεις απέναντι στην Τουρκία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουν όλες αυτές οι ιδεοπραγίες, να προχωρήσουμε προς ένα καθεστώς ειρήνης. Αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε την ειρήνευση ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους, δεν θα καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Η κατάσταση είναι σίγουρα πάρα πολύ ενισχυτική και όχι μόνο στην νότια-ανατολική Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έθιξε βέβαια η συγγήτρια, η κατάσταση δηλαδή όσο αναφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του τύπου. Πάλι εδώ πέρα σαφώς οπισθοδρομούμε. Δεν σημειώνεται πρόοδο στους τομείς αυτούς. Θα ήθελα πραγματικά μια μέρα να μπορούσαμε να είχαμε μια έκθεση για την Τουρκία που είναι λίγο πιο αισιόδοξη, που θα μπορούσε να ταινίσει το μέλλον με μεγαλύτερη φιλοδοξία και αισιοδοξία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σαφώς δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την επίλυση της προσφυγικής κρίσης με την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δεν μπορούμε επίσης να απομακρυνθούμε από τις βασικές μας θεμελιώδεις αξίες στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης αυτής, μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να κλείσει τα σύνορά της στους πρόσφυγες ε, η Τουρκία. Έχουμε θεμελιώδεις αξίες, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν, πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση και τα βασικά κριτήρια τα οποία θέτουμε απέναντι στην Τουρκία προκειμένου να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα θεμελιώδη κριτήρια, μόνο και μόνο επειδή θέλουμε την συνεργασία της Τουρκίας στο προσφυγικό ζήτημα. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις δύο πλευρές της διένεξης. Θα πρέπει και από τις δύο πλευρές να σταματήσουν οι βιοπραγίες. Να επικεντρωθούμε επίση στο γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Εμείς και η πολιτική ομάδα μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες συμβαστικές προτάσεις, ορισμένες λίγες δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Πάντως, πολλές φορές συμφωνούμε με την ουσία κάποιων συμβαστικών προτάσεων, όχι με την διατύπωσή τους. Ιδίω ε, δεν συμφωνούμε με τις τροπολογίες εκείνες που έχουν να κάνουν με την παράτυπη μετανάστευση. Δεν αναγνωρίζουμε την παράτυπη μετανάστευση, δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη μετανάστευση. Θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εγκαταλείψουν εμπόλεμε ζώνε και να ζητήσουν ειρήνη και μια ειρηνική ζωή αλλού στον κόσμο. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στους ε, υπόλοιπους ομιλητές. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ. Κύριο κύριος πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτριά μας, την κυρία Πύρη και τους κοιόδες εισηγητές. Και εγώ θέλω να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στα θύματα και τις οικογένειές τους μετά από αυτήν την άλλη μία τρομοκρατική επίθεση. Η Τουρκία είναι σημαντικό εταίρος της Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί και εταίρο κλειδί όχι μόνο για τη σταθερότητα στην περιοχή και την Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα όσον αφορά το προσφυγικό. Και αυτό είναι το leitmotiv αν θέλετε ολόκληρης αυτής της ιστορίας. Οι συνομιλίες, οι σχέσεις που έχουν τα διάφορα θεσμικά όργανα με την Τουρκία στρέφονται ακριβώς γύρω από αυτό. Η Τουρκία είναι επίσης μια χώρα η οποία πραγματεύεται για την ένταξή της. 3 Οκτωβρίου του 2005 άρχισαν αυτές όπως έγινε και με τη δικιά μου τη χώρα, πριν από 10 χρόνια δηλαδή η πρόοδος τα τελευταία χρόνια ήταν πολυμερική. Είμαι όμως πεπισμένος ότι πηγαίνοντας προς αυτή την κατεύθυνση και πιέζοντας περισσότερο για μεταρρυθμίσεις, κυρίως στο δικαστικό τομέα, το κράτος δικαίου, την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία έκφρασης, είναι στοιχείο κλειδί για την πρόοδο της Τουρκίας. Συνεπώς, οι συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες καταλήξαμε στέλνουν ένα πολύ καλό μήνυμα προς την Τουρκία αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή και ελπίζω να συμφωνήσετε με αυτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Παπαδάκης τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φετινή έκθεση απεικονίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα που ισχύει στην Τουρκία. Δυστυχώς Κάθε μέρα που περνάει έχουμε λιγότερη δημοκρατία στην Τουρκία, κάτι που κανείς από εμάς εδώ δεν θα το θέλαμε. Όσον αφορά τις αναφορές για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι αδιανόητο να λείπει αναφορά μέσα στην έκθεση ότι η λύση, η όποια λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι συμβατή με το κοινωτικό εγκεχτημένο και να στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας θα έπρεπε να ήταν θέμα αρχής. Και ξέρετε η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα το οικοδόμημα για τον λόγο ότι παραλείπουμε τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με τις παρεμβάσεις μας. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ και εγώ θέλω να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων μετά από αυτήν την δρομοκρατική επίθεση. Υπάρχουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίες έκφρασης με το κλείσιμο της εφημερίδας Ζαμάνα Υπάρχουν οι προειδοποίησει του Ερτογκάν όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο. Επίσης, οπολύθηκαν δύο δικαστές οι οποίοι αναφέρθηκαν σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ISIS, PKK κτλ. Η Τουρκία όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν άλλη λύση παρά να συζητάνε με την Τουρκία για να σταματήσει η εισρωή προσφύγων από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί και η διαδικασία ένταξης ή η κατάργηση των θεωρήσεων ή να μην συνεχιστεί η πίεση όσον αφορά το Κυπριακό. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουμε όλα αυτά αν προηγουμένως δεν εφαρμόσει η Τουρκία τα διάφορα πρωτόκολλα, διάφορες συμφωνίες της Άγκυρας κλπ. και αναγνωρίσει την Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος. Όμως το 2016 υπάρχει ελπίδα η Τουρκία να συμφωνήσει τελικά με μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και να ανοίξουν ίσως και τα σύνορα με την Αρμενία. Είναι μια δύσκολη έκθεση αυτή. Στη χώρα μου θα έχουμε το δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο όχι και τώρα μπαίνει το Κυπριακό στην συζήτηση αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ επίμαχο ζήτημα και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Κυπριακό δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αυτή η συζήτηση ε, βέβαια λαμβάνει χώρα σε μια ε, περίοδο όπου οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Τουρκία βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο και πραγματικά είναι μια σουρεαλιστική εμπειρία γιατί βλέπουμε τα όσα λαμβάνουν χώρα τώρα ουσιαστικά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την δεξιακή διαδικασία, την απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων, η έκθεση η οποία προέρχεται είχαν παγώσει για πάρα πολύ καιρό και ξαφνικά άρχισαν να ανακοινούνται όλα του. Και βέβαια βλέπουμε ότι ελπίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μαλακώσει τι αρχέ τη γιατί ελπίζοντας ότι δηλαδή θα μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματά της με την Τουρκία ε, ε, δεν ε, θέλουμε αυτό να επιληθεί δηλαδή εις βάρος των πολιτών. Κάτι τέτοιο θα αποβεί εις βάρος και ήδη αποβαίνει εις βάρος της αξιοπιστίας και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί δηλαδή πολίτες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Τουρκίας είναι πολύ απογοητευμένοι βλέποντας τα όσα συμβαίνουν και χαίρομαι πολύ ότι το Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή εστιάζουν σε αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα τα δικαιώματα των ανθρώπων και όλων των, των ανθρώπων, δηλαδή όχι μόνο των πολιτών της χώρας αλλά ε, και των ε, Κούρδων, των Κυρικών των ε, ανθρώπων LGBT και ούτω καθεξής. Αλλά και άλλες ελευθερίες όπως η ελευθερία του τύπου, του, διαδικτύου, της έκφρασης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να έχουμε την σωστό διαχωρισμό των εξουσιών και βέβαια ο έλεγχος της χρηστής διακυβέρνησης παραμένουν πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα θέσουμε προτού ολοκληρωθεί και παγιωθεί η συμφωνία που θα επιτευχθεί με την Τουρκία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να επιστήσω στην προσοχή σα σε κάτι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Αυτό που θα υπερασπιστώ τώρα είναι οι αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που οφείλει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόματα να εφαρμόσει στην έκθεση που αφορά την Τουρκία. Θεωρώ ότι η ενταξιακή πορεία τη Τουρκία δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπόθεση που αφορά πρωτίστω την Τουρκία. Η Κύπρο, να θυμίσω, τι 3 Δεκάτου του 2005, παρά το ότι βρισκόταν υποκατοχή, παρά το ότι παραβεζόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, έδωσε πράσινο φω στην Τουρκία για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υποσχέθηκε και δεσμεύτη να εφαρμόσει το πρωτόκολλο που ίδια υπέγραψε, όχι μόνο δεν το εφάρμοσε εδώ και 11 χρόνια, αλλά συνεχίζει να προκαλεί και να μην αναγνωρίζει χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω του αγαπητού συναδέλφου, εάν μια άλλη υποψήφια χώρα δεν αναγνώριζε τη χώρα του, εάν θα έδιναν το δικαίωμα ή τη δυνατότητα να ανοίξει οποιοδήποτε κεφάλαιο για την ενταξιακή πορεία. Άρα για μας δεν είναι κόκκινη γραμμή, αλλά τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να ανοίξει κεφάλαιο εάν η Τουρκία δεν υλοποιήσει τι υποχρεώσει. Και ένα άλλο τελευταίο. Κύριε Πρόεδρε, δόθηκε σε όλου 1,5 λεπτό, παρακαλώ, όπω μου εμένα. Είναι το θέμα των επίκων. Είναι ζήτημα έγκλημα πολέμου. Δεν μπορούμε εμεί σήμερα να λέμε ότι δεν στηρίζουμε την άποψη ότι πρέπει να αφαιρεθεί από την έκθεση το ζήτημα που έχει να κάνει με του έπικου και που χρεωτικά πρέπει να αφαιρεθούν. Και το δεύτερο και σημαντικό η λύση πρέπει να βασίζεται στι αρχέ και τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θεμελιώδε και πιστεύω ότι θα έχουμε την υποστήριξη όλων των συναδέλφων βουλευτών. Ο κύριο Μαυρίδη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εγώ θα, πραγματικά θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση ότι ο ανθρώπινο πόνο είναι παντού ο ίδιο και αυτό αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά στην τελευταία απώλεια ζωή που είχαμε στην Άγκυρα. Αλλά η απώλεια ζωή και ο ανθρώπινο πόνο είναι ο ίδιο και στι κουρδικέ περιοχέ, όπω ήταν και πριν μερικέ δεκαετίε στην Κύπρο. Έρχομαι τώρα στην έκθεση, καθ' αυτό έκθεση. Θα ρωτήσω του συναδέλφου εδώ, γιατί ήμασταν και πέρσι και κουβεντιάζαμε πάλι για την έκθεση προόδου τη Τουρκία. Τι πάει στραβά με την Τουρκία. Εγώ του απαντώ. Πάει στραβά εκείνο το οποίο είναι ω εξή συμφωνούμε συνεχώς πράγματα με την Τουρκία τα οποία δεν τα εφαρμόζει. Και φτάσαμε στο σήμερα. Έγινε ήδη αναφορά για άλλο κράτος μέλος μας το οποίο ξεκίνησε πριν 10 χρόνια ενταξιακές και είναι εντός. Η Τουρκία δεν είναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, τις αρχές και αξίες όπως λέχθηκε για την Κύπρο και όλα αυτά εμείς πρέπει να επιμένουμε, όχι να περιμένουμε κάποιους άλλους. Δύο τελευταίες κουβέντες. Ιούγκλος. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο προσχέδιο της έκθεσης, ούτε στην έκθεση για την Κύπρο. Το πρωτόκολλο 10, κύριε Πρόεδρε, κάνει αναφορά στο κοινοτικό ακτιμένο σε όλη την Κύπρο. Η Κύπρος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ούτε άλλο κράτος, ούτε constituent state. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Μαυρίδη. Λυπάμαι. Η κυρία Θεοχάρης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την έκθεση αυτή καταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία και στην πραγματικότητα γινόμαστε συνυπεύθυνοι για την λειτουργία ενός Ισλαμικού κράτους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς και ας αναλάβει τις ευθύνες του για αυτό το ζήτημα δεν αναφέρεται το, η έκθεση ούτε σε ένα λαό, ούτε, σε όλε, ούτε στις αρχές και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των οποίων θα πρέπει να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα, αλλά επιμένει να ονοματίζει μια λύση η οποία δεν θα γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό λαό και σας προειδοποιώ από τώρα να το ξέρετε, γιατί αυτή η λύση θα παραβιάζει τα δικαιώματα του κυπριακού λαού στο Επισημαίνω ότι στο πρωτόκολλο 10 με το οποίο εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο αναστέλλεται στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Εσείς μιλάτε αυτή τη στιγμή για νέο συνειδητικό κράτος, το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να επεκταθεί το κεκτημένο. Παραβιάζουμε τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ήδη ως, ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να πω πάρα πολλά για το Κυπριακό. Θα τελειώσω λέγοντα ότι η Τουρκία ε, για, να, ευχαριστήσω και τον συνάδελφο που μου έδωσε τον χρόνο, ε, θέλω να πω ότι η Τουρκία όσον αφορά το ζήτημα της ε, διοχέτευσης παρανόμως μεταναστών στην Ευρώπη δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υποστηρίζει τη μαφία εκείνη η οποία διοχετεύει τους, ε, τους καημένους τους πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. <laughs> Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την έκθεση αυτή, η οποία ο συνήθως είναι ισορροπημένη, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της κατάστασης στην Τουρκία. Πολλά τραγικά γεγονότα έχουν λάβει χώρα στην περιοχή αυτή, τα οποία μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Τα προβλήματα της Τουρκίας, ορισμένα τουλάχιστον από τα προβλήματα της Τουρκίας, είναι εσωτερικής φύσης, αλλά έχουν ε, εισαχθεί απ' έξω αν θέλετε. Η Τουρκία δεν είναι αυτή που ήταν πριν από δύο-τρία χρόνια. Εξακολουθεί και αποτελεί πάντως στρατηγικό μας εταίρο και πάντα θα μας ε, αφορά τελικά όσον αφορά τα οικονομικά μας συμφέροντα, την ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο στον τρόπο με τον οποίο συζητάμε ή επικρίνουμε πολλές φορές την Τουρκία. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ακόμα και οι δικέ μας συζητήσει μπορούν τελικά να επηρεάσουν την κατάσταση στην Τουρκία και νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε, να τοποθετούμε θα με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσαμε τελικά να ωφελήσουμε κάποιους ε, ακραίους πολιτικούς στην Τουρκία. Υπό το φως των εκλογών επίσης στην Γερμανία είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι ε, η ενσωμάτωση των Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία και σε άλλες χώρες ουδέποτε αποτέλεσε πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό το φαινόμενο και αυτή τη διαπίστωση θα πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Επιστελέγιος. Ο κύριος Επιτίδιος έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε εναντίον κάθε μορφής βίας και την καταδικάζουμε από πουδήποτε και αν προέρχεται. Υπό το πρίσμα αυτό καταδικάζουμε την ε, ενέργεια, την τρομοκρατική που έγινε πρόσφατα στην Άγκυρα και είχε θύματα δυστυχώς μόνο ανθρώπους ανθρώπους, στους συγγενείς των οποίων ειλικρινά συλληπούμε. Δυστυχώς η βία είναι μια εγγενής αδυναμία του τουρκικού κράτους και την εφαρμόζει κυρίως απέναντι στους δικούς του πολίτες. Επίσης, έχει μια επιθετική πολιτική η Τουρκία απέναντι στους γείτονές της. Ξέρετε όλοι ότι απειλεί την Ελλάδα με κάζους Μπέλη, δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία τη οποία κατέχει παράνομα το 38% του εδάφους, έχει, το έχει επικίσει, προσπαθεί να λιώσει την πληθυσμιακή του σύνθεση και σε κάθε περίπτωση είναι επιθετική. Αυτή τη χώρα την έχουμε αναβαθμίσει ως ισότιμο συνομιλητή σε θέματα επιλύσεως του προσφυγικού. Δυστυχώ δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκβιάζει και δεν πρέπει να ανεχθούμε μια τέτοια κατάσταση. Τέλο, θέλω να πω το εξή. Εάν υπάρχει ένα λαό ο οποίο οφείλει να δεχτεί τα συγχαρητήριά μα, αυτό είναι ο ελληνικό λαό, ο οποίο εξουθενόμενο από τα μέτρα του μνημονίου, ανέχεται ακόμη την κυβέρνησή του να δέχεται και να εγκαθιστά στη χώρα όλου αυτού του παράνομου μετανάστε. Αντιθέτω, η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτού του δυστυχεί ανθρώπου και κερδοσκοπεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπροκ, τελευταίος. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, συγγύτρια Κατυπηρή και τους υπόλοιπους σκιώδεις συζητητές ε, για ένα σχέδιο έκθεση το οποίο πραγματικά είναι ισορροπημένο. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποια, κάποιες βασικές παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά την ε, Τουρκία. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία του τύπου, ελευθερία της έκφρασης και άλλες ελευθερίες και γνωρίζουμε πως αυτός ο πόλεμος κατά των Κούρδων είναι αχρίαστος και αποτελεί πραγματικά ένα πολιτικό μέσο που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα η Τουρκία και αρχίζει να γίνεται ανεξέλεγκτο. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι συμβαίνει με κάποια κράτη-μέλη ε, τα οποία τώρα τάσσονται ενεργά κατά της προσχώρησης της, Τουρκία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ήταν πολύ ανοιχτά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Όταν εγώ τότε ήδη είχα ευστήσει την προσοχή στα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία παρά την κριτική που της ασκούμε αποτελεί ακόμα σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον μια δημοκρατία εάν τη συγκρίνουμε δηλαδή με την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Ε, δηλαδή όλες οι υπόλοιπε μουσουμαλικές χώρες ε, γύρω από την Τουρκία ε, βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την Κύπρο. Για πρώτη φορά δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει, να διακρίνεται μία πολύ σαφή ευκαιρία για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια επίλυση για το κυπριακό ζήτημα με υψηλό βαθμό σοβαρότητας και από τις δύο πλευρές. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, ναι, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε μια τέτοια λύση. Ε, και εγώ θεωρώ πως ο πρόεδρος της ε, Κυπρίας της Δημοκρατίας με την πρόταση που έκανε σε ό,τι αφορά την ε, τουρκική γλώσσα, αποτελεί πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ιδέα γιατί θα μπορούσε ενδεχομένω να βοηθήσει στην ε, διαδικασία συμφιλίωση. Και θεωρώ πως βέβαια πολύ σημαντικό το γεγονό ότι αυτή η πρόταση προήλθε από την πλευρά του Πρόεδρου τη Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει ε, να παραμείνουμε απλά ε, στα όσα έχουμε, υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε ε, κάτι, να υπάρξει μια δυναμική στη διαδικασία για να μην είμαστε σε 20-30 χρόνια στην διακατάσταση. Και α μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία παίζει εδώ ένα σημαντικό ρόλο. Αν θέλουμε δηλαδή ο αριθμός των προσφύγων να μειωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν επιθυμούμε να μείνουν όλοι παγιδευμένοι οι πρόσφυγες στην Ελλάδα αφού κλείνουν όλες οι υπόλοιπε ε, οδοί και βέβαια είμαι κατά αυτού του κλεισίματος ε, της ε, οδού των Βαλκανίων θα καταλήξουμε με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούν και οι φίλοι μας από την Ελλάδα τι θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή θα συνεχίσουν να έρχονται οι πρόσφυγες από την Τουρκία, δεν θα υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν κλείσει και τα σύνορα. Τι θα γίνει, θα είναι έξυπνη μια τέτοια λύση. λύση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω, παρά την κριτική που ασκούμε και την οποία κατανοώ βέβαια, ε, γιατί προέρχεται και από ιστορικούς λόγους, να λάβουμε και αυτά τα ζητήματα υπόψη μας. Σε ό,τι αφορά ε, την ενταξιακή διαδικασία. Χρειαζόμαστε 72 καταρχήν ε, ε, ε, ομόφωνε σε επίπεδο κρατών μελών για να πούμε ότι θα μπορέσει να προσχωρήσει ένα νέο κράτος μέλος. Σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια και τα ανοίγματα, ακόμα είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμός των κεφαλαίων που έχουν ανοιχθεί. Οπότε πραγματικά δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση κοντά σε μια ένταξη της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό βρίσκεται ακόμα μακριά. Μετά σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτος ε, των θεωρήσεων, ναι, προφανώ εδώ θα πρέπει να ε, θίξουμε και αυτά τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διαφόρων ελευθεριών. Θα πρέπει δηλαδή να πρέπει να υπάρξει ένα πολύ αυστηρό έλεγχο αυτών των ζητημάτων για να καταστήσουμε σαφέ ότι η Τουρκία δεν ε, είναι έτοιμη για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό θα πρέπει να τεθεί και στο πλαίσιο του διαλόγου σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων. Η διαπραγμάτευση δηλαδή που θα γίνει σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων θα πρέπει να ακολουθήσει την διαπραγματευτική διαδικασία που ακολουθούμε και σε ό,τι σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, σε όλε τι υπόλοιπε διαπραγματεύσει. Σα είπα λοιπόν, 72 κριτήρια έχουμε συνολικά που θα πρέπει να τηρεί και 72 συμφωνίε, αλλά δεν ε, ε, τηρείται ένα πολύ μεγάλο αριθμό και ε, δεν μπορούμε να κάνουμε πτώσει σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, για να μπορεί να πληρεί αυτά τα 72 κριτήρια θα πρέπει να έχει επιτύχει και τις κατάλληλε ε, πρόοδου σε ε, πολιτικό επίπεδο η Τουρκία και γι' αυτό ακριβώ θεωρώ το πως ε, η έκθεση κινείται προς τη κατή κατεύθυνση και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά την εισηγήτα κυρία Πύρη. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόκ. Η κυρία Πύρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν περίμενα ότι θα έφτανε σε μένα ο λόγος και πάλι Γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των πολιτικών ομάδων κάθε φορά που συζητάμε για την Τουρκία. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση και μετά την ανάλυση που έχουμε κάνει όλες οι μεγάλες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε κάποια συμφωνία. Υπάρχει κάποια ανησυχία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την έκθεση για την Τουρκία εδώ στην αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει έλεγα Πρόεδρε, ότι σήμερα το απόγευμα μπορούμε γρήγορα να ψηφίσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και το σύνολο της έκθεσης. Και μετά στην Ολομέλεια τον Απρίλιο στο Στρασβούργο θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε κυρία Πύρη. Όντως στις 4 θα ψηφίσουμε. Τελειώσαμε με αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το, της Μέρης συγγνώμη. για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Silent, please. Vamos a Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, παρακαλώ. Καλωσορίζω εδώ τον Γέρση Πιομανόφσκι, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του Ταμείου αυτού, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 2013 λειτουργεί πλήρως και έχει δραστηριοποιηθεί όλος ιδιαίτερος αυτά τα τρία χρόνια που λειτουργεί. Δημιουργήθηκε μετά από κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών και βασίζεται στο βελγικό δίκαιο. Έχει αναλάβει ήδη 150 πρωτοβουλίες και το 2015 θέλησε να επεκταθεί περισσότερο και να μην μείνει μόνο στις γειτονές χώρες. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πομιανόφσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Με ιδιαίτερη περηφάνεια θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητές μας για το 2015 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Ξέρω ότι στα πλαίσια του καταστατικού του Ταμείου αυτού οφείλω να έρχομαι εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας παρουσιάζω τις δραστηριότητές μας. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν βρίσκομαι σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες αυτές. Υπάρχει μια ηλεκτρονική εκδοχή Τη έκθεση αυτή και έχουμε φέρει και κάποια έντυπα αντίγραφα τη έκθεση τα οποία μπορούμε να διανύμουμε σε εσά εφόσον το επιθυμείτε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια κέρια σημεία της δραστηριότητάς μας και στη συνέχεια βέβαια είμαι στη διαθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία κατά το 2015, μια δραστηριότητα η οποία ξεπέρασε τις βασικές δραστηριότητες του EED και αναφέρουμε αυτή τη στιγμή σε μια δική έκθεση όσον αφορά τη ρωσική γλώσσα και τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Ρωσία, μαζί της συγκεκριμένη κυβέρνηση της Ολλανδίας να ασχοληθούμε με το ζήτημα της ρωσικής προπαγάνδας, ιδίως στα πλαίσια της αντολικής εταιρικής σχέσης, που ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους στην περιοχή αυτήν. Να αναφερθώ επίσης στη γεωγραφική επέκταση του EED, προκειμένου να καλύψουμε και τους γείτονες των γειτόνων μας, απόφαση που ελήφθη στα τέλη του 2013 και άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από το 2015. Τέλος, θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία δίνοντάς σας κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και σκιαγραφώντας γενικότερα τα όσα έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όσον αφορά την ρωσική γλώσσα και τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατά έξι μήνες του 2015 κάναμε λοιπόν μία έρευνα, δημοσιεύσαμε την έκθεση αυτή η οποία είχε ως στόχο να συμπεριλάβει τις χώρες εκείνες που ενδιαφέρονταν για την έκβαση αυτής της μελέτης. Πρόκειται για μια μελέτη ε, σκοπιμότητος που είχε ως βασικό στόχο να απαντήσει στο εξής ερώτημα. Πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε την επιρροή του Κρεμλίνου και γενικότερα του ρωσικού κράτους όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκπέμπουν στη ρωσική γλώσσα. Ξέρετε ότι ε, πρόκειται ουσιαστικά για τα μέσα εκείνα τα οποία επηρεάζει το Κρεμλίνο προκειμένου να προωθεί την προπαγάνδα του προ ένα ευρύτερο κοινό και ακροατήριο. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που θέσαμε είναι αν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα νέο μεγάλο ευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμίσει κάπως την προπαγάνδα που κάνει η ρωσική πλευρά. Προσπαθήσαμε πάντως για την έβρεση μιας συγκεκριμένη λύσης να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε ως Ευρωπαίοι με τρόπο πάρα πολύ συντονισμένο και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας και τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν και για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει ένας περιφερειακός συντονισμός. Θα πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα νέο τηλεοπτικό κανάλι αυτό ήδη απαντάται από τον τίτλο της ε, έκθεσης όπου λέμε ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε τον πλουραλισμό και την εξαρτησία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ρωσίας. Ιδιαίτερη αναγνώριση έλαβε η έκθεση αυτή. Αναφέρθηκε επίσης σε πάρα πολλά ρεπορτάζ που κάνανε δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και επίσης ε, αναφέρθηκε στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την ανατολική εταιρική σχέση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και επίση, πάρα πολλέ κυβερνήσει σε διάφορε συνδιασκέψει που έγιναν μετά την έκθεση αυτή λάβαν υπόψη του τις συστάσει που γίνονται σε αυτή την έκθεση και έχουν πει ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τις συστάσεις της έκθεσης αυτής στα προγράμματα εξωτερική πολιτική και στην κατανομή πόρων εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Η δημιουργία ανεξάρτητων λοιπόν μέσων μαζική ενημέρωση ω πρώτη σύσταση το ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο αριστείας μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα αναλύει τις γενικότερες τάσεις και την κατάρτιση των δημοσιογράφων στην ευρύτερη αυτή περιοχή και που κατά αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσει στο να έχουμε ανεξάρτητες ειδήσει στην περιοχή αυτή. Οι τρεις αυτές συστάσεις πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν και υπάρχει ακόμα μια τέταρτη σύσταση η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ορισμένους μήνες λοιπόν μετά την δημοσίευση της έκθεσης αυτής έχουμε τρεις συστάσεις τις οποίες έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του χώρες όπως οι κάτω χώρες, το Μένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Αυτά όσον αφορά τη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία εκεί πέρα που χρειάστηκε δηλαδή να υπερβούμε τη βασική μας κεντρική εντολή και όπου τελικά κάναμε μια πολύ ειδικευμένη εργασία που είχε να κάνει με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το οποίο είπαμε ότι θα πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένες συστάσεις και δράσεις. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι στα πλαίσια των κεντρικών μας δραστηριοτήτων το 1 τρίτο των έργων μας στην περιοχή έχουν, έχει να κάνει με την υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Το 1 τρίτο λοιπόν των σχεδίων μας, των έργων μας, ήδη υποστηρίζουν τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα με το αν έχει συνταχθεί για αυτά έκθεση ή όχι. Δεύτερον, όσον αφορά την γεωγραφική επέκταση της εντολής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη σε μια συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, Δεκέμβριος του 2014. Η διαδικασία εφαρμογής ξεκίνησε ήδη από το 2015. Και βέβαια συνειδητοποίησαμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε κάπως τη δράση μας γιατί είναι περιορισμένοι και οι πόροι μας καθώς επίσης και τα χρηματοδοτικά κονδύλια. Το Συμβούλιο αποφάσισε λοιπόν ότι θα πρέπει να επεκταθεί η γεωγραφική μας κάλυψη αλλά δυστυχώς αυτό δεν συνοδεύτηκε με, με την απαραίτητη αύξηση της χρηματοδότησής μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ως ε, γραμματεία θα πρέπει να καταφέρουμε να συντονιστούμε και με την εκτελεστική μας επιτροπή και με το Συμβούλιο και θα πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να καταφέρουμε να υπερβούμε την αρχική γεωγραφική μας εντολή που κάλυπτε μόνο την νότια και ανατολική γειτονία. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να επικεντρωνόμαστε πλέον σε κάποιες ε, περιοχές για τις οποίες είτε δίνουν χρηματοδότηση τα μέλη μας, είτε θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ορισμένα σχέδια, ορισμένα έργα είχαν να κάνουν με εταίρους μας στην Ρωσία και γενικότερα στην Κεντρική Ασία. Επίσης ε, ξεπεράσαμε την ε, ευρύτερη γειτονία μας και πήγαμε ακόμα και μέχρι τα αραβικά κράτη. Ασχοληθήκαμε με τον Μπαχρέιν. Πάντως στα πλαίσια του 2015 δεν ελήφθησαν κάποιες σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τις περιοχές αυτές. Κινούμεθα περισσότερο σταδιακά και βαθμία για να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε και άλλες περιοχές. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε περισσότερους δωρητές και προσπαθούμε, όπως σας είπα, να υπερβούμε την κλασική μας, τη συνηθισμένη γεωγραφική μας κάλυψη. Προκειμένου βέβαια να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και να υπερβούμε την αρχική μας γεωγραφική εντολή θα καταστεί δυνατό μόνο όταν καταφέρουμε να έχουμε επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους. Και να πω ορισμένα πράγματα και για τις ε, βασικές μας δραστηριότητες και να δώσω κάποια παραδείγματα. Το 2015 είχαμε πλέον δύο πλήρη έτη πλήρους δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Καταφέρνουμε και υποστηρίζουμε λοιπόν τη δημοκρατία και τον εκδημοκρατισμό και ακόμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει πλέον τη δράση μας. Αυτό φάνηκε άλλωστε στην έκθεση που ψηφίσατε τον Ιούλιο. Ο σημαντικό μα ρόλο επίση αναγνωρίζεται και στην υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών στα πλαίσια τη ε, αναθεώρηση ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, όπου συμβάλαμε κι εμεί μέσω των εταίρων μας. Think tanks όπως το Carnegie Europe έχουν αναγνωρίσει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία συμβάλλει πάρα πολύ σε συγκεκριμένε δράσεις εκδημοκρατισμού και αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο και εξόλογο εταίρο όσον αφορά την υποστήριξη για τη δημοκρατία. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία καταφέρνει πλέον και συμπληρώνει την δράση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων δωρητών. Στην πράξη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία καταφέρνει και έχει πολύ σημαντική υποστήριξη σε ορισμένες χώρες όπου πρέπει να ληφθεί επιγόντως δράση, όπως να υποστηρίξουμε για παράδειγμα την ε, κοινωνία των πολιτών στην Αρμενία με, πριν το δημοψήφισμα το οποίο έγινε για να τροποποιηθεί το σύνταγμα της χώρας. Ορισμένοι δωρητές χορηγοί μας δεν κατάφεραν να αποκριθούν όσο γρήγορα αποκριθήκαμε εμείς. Επίσης η προστιθέμενη αξία μας φαίνεται στο ότι συμβάλλουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα από πολιτικής πλευράς και τα οποία δεν καλύπτονται στα πλαίσια διμερών σχέσεων. Υποστήριξη δηλαδή Αντιπολίτευση η Μολδαβία και η Ουκρανία, όπου στόχος μας εκεί πέρα να καταφέρουμε να δώσουμε στους ψηφοφόρου μια εναλλακτική δημοκρατική επιλογή για το μέλλον. Επίσης πολλές φορές παίρνουμε ε, ρίσκα και καταφέρνουμε και υποστηρίζουμε νέε δημοκρατικέ ομάδε σε κάποιε χώρε, οι οποίε δεν έχουν την υποστήριξη συγκεκριμένων δωρητών, όπω ε, το Μαϊντάν στην Ουκρανία, ένα κίνημα το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά μετά την ε, δημιουργία της, ε, του βασικού κινήματος Μαϊντάν στην Ουκρανία. Από την αρχική αυτή ομάδα δημιουργήθηκε μια επιμέρους ομάδα ακτιβιστών που χρησιμοποιεί οχήματα, αυτοκίνητα, κάνει περιοδία στη χώρα και προσπαθεί να ταχθεί κατά της διαφθοράς της αστυνομίας. Είχαν μια αρχική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και αφού γίνανε γνωστοί χάρη σε εμάς, κατάφεραν να προσελγίσουν μια ευρύτερη υποστήριξη προκειμένου να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα διαφθοράς στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια ή σε διάφορες εθνικές αρχές όπως οι αστυνομικές αρχές κτλ. Χρησιμοποιούν επίσης διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλές φορές ανεβάζουν βίντεο τους σε εφαρμογές όπως το YouTube και σε άλλες εφαρμογές. Επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία υποστήριξε στην Μολδαβία δύο websites, Newsmaker και Wall Street, που ε, ουσιαστικά αναφέρθηκαν στην ε, διαφθορά της κυβερνητικής ελίτες σε αυτή την υπεξαίρεση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που είχε να κάνει με το τραπεζικό σκάνδαλο της χώρας. Προσπαθήσουμε επίσης να υποστηρίξουμε τους εταίρους μας οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πολύ δύσκολες εμπόλεμες ζώνες όπως η Συρία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία προσπαθεί να προωθήσει τον εκδημοκρατισμό της Συρίας, βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας των πολιτών και προσπαθεί να ενθαρρύνει το κράτος δικαίου, την ελευθερία του τύπου και τον διακοινωτικό διάλογο. Επίσης προσπαθούμε να υποστηρίξουμε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Στο Αζερβαϊτζάν και στην Αίγυπτο έχει δεικνωθεί πάρα πολύ ο χώρος δράσης της κοινωνίας των πολιτών και προσπαθούμε και εκεί ως Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία να υποστηρίξουμε τις φιλοδημοκρατικές ομάδες των χωρών αυτών, ότι το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα αντίξω σε, στα πλαίσια εχθρικών ε, περιβαλλόντων, εχθρικών ε, περιοχών. Προσπαθούμε ως Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Δημοκρατία να προωθήσουμε τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης. Να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε δηλαδή όλους εκείνους ακτιβιστές που διακινδυνεύουν πολλές φορές και τη ζωή τους προκειμένου να προωθήσουν και να προασπίσουν τις αρχές τους. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των ακτιβιστών και να τους υποστηρίξουμε συμπεριλαμβανομένης πολλές φορές ακόμα και της προστασίας της ίδιας τους της ε, ταυτότητας. Θα σας δώσω τώρα κάποια αριθμητικά δεδομένα. Το 2015 το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία χρηματοδότησε 114 νέες πρωτοβουλίες, 19 εκ των οποίων είχαν να κάνουν με νέες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 842 αιτήσει για υποστήριξη έχουμε λάβει. Και έχουμε εγκρίνει 10 με 12% από αυτές. Επίσης, Κάναμε 112 επισκέψεις παρακολούθησης σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες δικαιούχους. Αυτό έχει γίνει μόνο με τα 16 άτομα τα οποία εκπροσωπούν 14 διαφορετικές χώρες που ουσιαστικά συνιστούν τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Όλα αυτά δεν θα είχαν όμως καταστεί δυνατά αν δεν είχαμε αποτελεσματικές ε, δομές διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Έχουμε 13 χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, την Εκκληστική Επιτροπή που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις χρηματοδότησης, αλλά και την πολύ ουσιαστική συμβολή από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αναφέρομαι μόνο στα εννέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, αλλά και σε όλου του υπόλοιπου ευρωβουλευτέ που συμμετέχουν με τον άλλο τρόπο στη δραστηριοποίηση του Ταμείου αυτού. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πομιανόφσκι. Πρώτον, θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Ο κύριος Μπρόκ, για παράδειγμα. Όχι. Όχι. Ο Αντρέσι τότε έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Πονιανόφσκι με ικανοποιούν. Διότι στην πραγματικότητα δείχνουν ακριβώς αυτά που περιλαμβάνονται και στην έκθεση την οποία συζητήσαμε ήδη. Η ετήσια αυτή έκθεση αναφέρει όλες τις πρωτοβουλίες, όλες τις δράσεις του Ταμείου αυτού για τη Δημοκρατία και αναφέρονται και λεπτομερώς και τα οικονομικά ζητήματα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκτελεστικό διευθυντή που ήρθε και μας συνόψισε την κατάσταση της δραστηριότητε του Ταμείου αυτού που συνάδουν απόλυτα με το περιεχόμενο της έκθεσης. 273 διαφορετικές πρωτοβουλίες έτυχαν στήριξη από το Ταμείο, από ό,τι φαίνεται. Πρόκειται για χώρες της γειτονίας όπως η Ρωσία, η ε, Βελορουσία, όπως η Αίγυπτος. Συνεπώς, διαπιστώνουμε κι εμείς να υπάρχει μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στις χώρες που γειτονεύουν άμεσα και σε εκείνες που βρίσκονται πιο μακριά. Αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν που στηρίχτηκαν προχώρησαν σε χώρες που γειτονεύουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτή η γεωγραφική επέκταση είναι πλέον ένα γεγονός. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι το Ταμείο λειτουργεί κάτω από όλο και πιο δύσκολες συνθήκες. Και γιατί, διότι οι δράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα και σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, κάτι το οποίο δεν διευκολύνει βέβαια το έργο του Ταμείου. Παρ' όλα αυτά, το Ταμείο βρίσκει πάντα έξυπνες ιδέες και νέες μορφές δραστηριοτήτων. Υπογραμμίζω επίσης και τη συνεισφορά των κάτω χωρών αναφέρθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής στη στήριξη των κάτω χωρών στις διάφορες δραστηριότητες του Ταμείου και στην καταπολέμηση της μασικής της υπερβολικής προπαγάνδας από πλευράς της Ρωσίας. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά και τις πηγές χρηματοδότησης, εννοείται ότι υπάρχουν κοινοτικές πηγές ανάμεσα σε δύο δόσεις, όμως συχνά υπάρχει ένα κενό. Οπότε πρόκειται για μια στήριξη η οποία είναι τακτική αλλά δεν είναι συνεχής. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στο Ολλανδικό σχέδιο, το οποίο ανέφερε και ο ίδιος εκτελεστικός διευθυντής. Η εμπειρία αυτή θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν λέω με κοινοτική χρηματοδότηση οπωσδήποτε, αλλά ίσως βρίσκοντας άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί, να επεκταθεί. Και μια που είμαι στο οικονομικό σκέλος, θέλω να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, ότι η Νορβηγία συμμετέχει τώρα στην ομάδα δωρητών. Και ο Καναδάς δέχτηκε να στηρίξει ένα σχέδιο που έχει να κάνει με την Ουκρανία. Αναρωτιέμαι λοιπόν το εξή. Προκειμένου να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα μια σταθερή χρηματοδότηση, δεν θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει μια διεθνή συμφωνία η οποία να υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο ή τέλο πάντων αναφέρει τις υποχρεώσεις των χωρών προκειμένου να στηρίζουν το ταμείο αυτό. Επίσης δεν είναι δυνατόν να μην μιλήσουμε και για τον αριθμό του προσωπικού. Δεν θα μπορούσαν να αποσπαστούν οι υπάλληλοι από τις χώρες μέλη που συμμετέχουν και να πάνε στο Ταμείο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό για το Ταμείο. Έπειτα, οι χώρες μέλη που έχουν ειδικευτεί κατά κάποιο τρόπο στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιείται το Ταμείο, ε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και πηγή προσωπικού για το Ταμείο αυτό. Ακριβώς επειδή είναι ειδική πλέον. Έτσι θα μπορούσε να υποφεληθεί το Ταμείο. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα λοιπόν για το προσωπικό και τέλος να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Διευθυντή αλλά και όλους τους συνεργάτες του που τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παντσέρη θα είμαι σύντομο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Πομανιώσκη για την εξαιρετική αυτή εργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Νομίζω ότι μας περιέγραψε την δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία με τρόπο απόλυτα σωστό και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στις αρχικές μας προσδοκίες αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Ξέρετε ότι ε, είχαμε συζητήσει τότε και έναν ε, προληπτικό προπολογισμό για το Ταμείο αυτό. Ιδίω ε, όσον αφορά τη δράση του στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Καταφέραμε, θεωρώ, να πετύχουμε την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στις πολιτικές υποστήριξης της νότιας και της ανατολικής γειτονίας αλλά όπως ακούσαμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία έχει αυξήσει την γεωγραφική του κάλυψη. Όλα αυτά αποτελούν θετικά στοιχεία στην αξιολόγηση του Ταμείου, συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν προβλήματα πόρων και χρηματοδότησης. Μία πρόταση που θα μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή ενώπιον του Διευθυντή και μέσω της συζήτησης που είχαμε κάνει στο παρελθόν πέρα από την ισορροπία αυτή που πετύχαμε σε επίπεδο πολιτικής, θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να επενδύσουμε κατά προτεραιότητα βάσει της επικαιρότητα της πολιτικής που ζούμε αυτή τη στιγμή. Πέρα από το ζήτημα της Ουκρανίας, νομίζω ότι ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα, στην νότια τουλάχιστον Ευρώπη, είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που έχουμε σε χώρες όπως η Τινησία και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε την σταθεροποίηση σε τέτοιες χώρες και να κάνουμε και επενδύσεις προς τις χώρες αυτές. Τέλος, υπάρχει και ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο είχαμε θέσει και στο παρελθόν, αποτέλεσε αντικείμενο και μια τηλεφωνική συνδιάλεξης που είχαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, που έχει να κάνει με την διεύρυνση της ε, χρηματοδοτικής εισφοράς πολλών χωρών προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό και η Ιταλία να μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί αυτό το ταμείο και νομίζω ότι δημιουργούνται πλέον πιο ευνοϊκέ συνθήκε προκειμένου να συμμετέχουν όλο και περισσότερε χώρε στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Αποτιμώ λοιπόν πολύ θετικά τη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Το τονίζω αυτό, αναγνωρίζω τη σημαντική συμβολή σα και τον εξαιρετικό ρόλο που διδραματίζει ο κύριο Πομανιώσκη. Ευχαριστούμε κύριε Παντσέρο. Κύριος Λάμστορφ έχει τώρα το λόγο. Yeah. Ευχαριστώ πολύ εγώ θα είμαι σύντομο στη δική μου παρέμβαση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Γομιανόφσκι ε, για αυτή την έκθεση. Θεωρούμε πως ε, αυτή η ετήσια έκθεση ε, στη γραπτή της μορφή πραγματικά επιτυχημένη και υπάρχουν και κάποια, κάποιες πτυχές που θα πρέπει να τις τονίσουμε από πολιτικής άποψη, δηλαδή ότι συνεργαζόμαστε ε, με το ε, Ταμείο εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή μια, ε, ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε καταρχήν την συνέχεια σε ό,τι αφορά το προσωπικό του Ταμείου, δηλαδή συνεχίζουμε και με τη δεύτερη περίοδο με, τον, με το ίδιο διοικητικό προσωπικό, δηλαδή με τον ίδιο ε, σύμβουλο και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε μια σταθερότητα για να αξιολογήσουμε τα πρώτα όσα επιτεύχθηκαν στην διάρκεια του πρώτου κύκλου. Ε, μια δεύτερη σημαντική πτυχή είναι ε, κάτι που ανέφερε και ο ίδιος ο κ. Σεπομιανόφσκι, ότι δηλαδή έχουμε μια διευρυμένη γεωγραφική εντολή. Δηλαδή αρχικά στο καταστατικό ε, η αναφορά που γινόταν έχει διαγραφεί, η αναφορά δηλαδή που γινόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τεμείου. Ε, και αυτή η διευρυμένη λοιπόν εντολή δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερα ασύνηθες, αλλά προφανώς συνεπάγεται περισσότερο φόρτο εργασίας για το προσωπικό του ταμείο. Οπότε χρειάζονται και περισσότεροι πόροι από την πλευρά των ε, κρατών μελών για να μπορεί να ανταποκριθεί το ταμείο στις υποχρεώσεις του. Οπότε απευθύνω και εδώ έγκληση προς τα κράτη-μέλη να υποστηρίξει το ταμείο με την διάθεση ε, περισσότερου προσωπικού. Αρχικά η κατάσταση ήταν ότι ή όπως είχαν οργανωθεί τα πράγματα, τα κράτη-μέλη ήθελαν να προβούν σε αποσπάσεις ε, ειδικών ε, από την πλευρά τους, όμως αυτό δεν συνέβη μέχρι στιγμής, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, στο μέλλον. Πάντως χαίρομαι που είναι πολύ ευρία η συνένεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τα όσα έχει επιτύχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Δημοκρατία και ε, βλέπω πως ε, η πλειοψηφία των ε, πολιτικών ομάδων υποστηρίζει εμφατικά τις εργασίες αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Θεωρούμε και εμείς λοιπόν ότι πραγματικά συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση των βασικών αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε Αστροβίτσιος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κύριο Πομιανόφσκι και την ομάδα του συγχαρητήρια για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής όσον αφορά τις δραστηριότητε του Ταμείου για το 2015. Αυτά τα οποία ε, κάνει, έχει εντολή να κάνει το Ταμείο, είναι στήριξη σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή γειτονίας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χώρος αυτός δεν βρίσκεται απαραίτητα σε ειρήνη. Ούτε υπάρχουν μόνο θετικές τάσεις. Βλέπουμε αποτυχημένες χώρες, βλέπουμε περιορισμό της δημοκρατίας, δύσκολες οικονομικές καταστάσεις σε πολλές χώρες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία λοιπόν έχει ένα μοναδικό πολιτικό προφίλ. Δραστηριοποιείται η διαπρωτοβουλία και έχει δραστηριότητες με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ των άμεσων γειτόνων μας. Θέλω να χαιρετήσω λοιπόν την δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία όσον αφορά την έκθεση σκοπιμότητας για την ρωσική γλώσσα και τα ρωσικά μέσα ήταν μία έκθεση που έκανε τη διαφορά όσον αφορά την κατανόησή μας πριν και μετά για τη ρωσική προπαγάνδα και τις ενημερωτικές δραστηριότητες. Αν δείτε λοιπόν το αποτέλεσμα γιατί είναι ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έκθεση σκοπιμότητας. Βλέπετε ότι η εξωτερική δράση και η Επιτροπή επικεντρώνονται τώρα σε τέτοιες δραστηριότητες, κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το ποια πρέπει να είναι η σωστή απάντησή μας όταν βλέπουμε να υπάρχει τέτοια προπαγάνδα και ένας πόλεμος ενημέρωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Είναι πολύ αποτητικό το έργο. Και υπάρχει και ανταγωνισμός όσον αφορά τους πόρους, δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Όμως, οι 114 πρωτοβουλίες που χρηματοδοτήθηκαν το 2015 σίγουρα θα βοηθήσουν να ενισχυθεί το προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θα επιτευχθούν και πολλοί από τους στόχους μας. Η ερώτησή μου τώρα προς τον κύριο Πομιανόφσκι έχει να κάνει με την συνεργασία του Ταμείου με το δίκτυο εταίρων στις γείτονες χώρες, που είναι σημαντικό πιστεύω για να καταλάβουμε τις ανάγκες και την κατάσταση ακριβώς. Πώς βλέπετε λοιπόν τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να επενδύσουμε πιο συγκεκριμένα και έπειτα η ιδιωσιμότητα των διαφόρων προγραμμάτων που έχουν στηριχτεί μέχρι τώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία το 2014 και 2015. Σε τι βαθμό δηλαδή τα χρήματα τα οποία δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο βοηθάει ώστε να υπάρξει κάποια διαφορά. Στα προγράμματα δηλαδή που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα σας και κάθε επιτυχία για το μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κομιανόφσκι, και εγώ ως Ευρωβουλευτής από την Ενωτική Αριστερά θέλω να σχολιάσω κάτι. Εμάς δεν μας ικανοποιούν τέτοιου είδους μέσα όπως αυτό το ταμείο. Το έχουμε ξαναπεί. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι ένα κακό αντίγραφο του κάθε εθνικού αντίστοιχου ταμείου για τη δημοκρατία. Σημασία έχει πώς χρησιμοποιείται ε, κάθε τέτοιο ταμείο που πολλές φορές πλήττει την κυριαρχία ακόμα και το ρόλο του ΟΗΕ με το άλλο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε εδώ για την ρωσική προπαγάνδα. Γιατί η ρωσική προπαγάνδα, δεν υπάρχει και άλλη προπαγάνδα. Υπάρχει και το CNN και αυτό κάνει προπαγάνδα. Οπότε, εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια επιτροπή που αποφασίζει τι είναι δημοσιογραφία και τι είναι προπαγάνδα. Εγώ νομίζω ότι το αντίβαρο πρέπει να έρθει αλλιώς, να υπάρξει πραγματικός πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει, υπάρχει το Russia Today, υπάρχει το Euronews, υπάρχει το CNN, υπάρχει και το Fox. Έτσι, η δικιά μου πολιτική ομάδα αυτό φοβάται, ότι και αυτά κάνουν προπαγάνδα. Αυτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ποβιανόφσκι για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις που απευθύνατε. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω το ταχύτερο δυνατό, αλλά όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Ξύπ για το γεγονός ότι έθεσε το ζήτημα σε μια μια ευρύτερη προοπτική, δηλαδή όχι μόνο την έκθεση του 2015, αλλά ε, στο πλαίσιο δηλαδή της ε, έκθεσης ε, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά δηλαδή την αξιολόγηση των δύο πρώτων ετών λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Και αυτή βέβαια η δική μας έκθεση τώρα για το 2015 αποτελεί και τη γέφυρα με αυτή την αξιολόγηση των πρώτων δύο ετών. Εμείς λοιπόν παρακολουθήσαμε από κοντά και σεβαστήκαμε ε, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες ε, γραμμές που λάβαμε, δηλαδή να παρακολουθούμε ε, από κοντά τόσο τους εταίρους μας από, την, από την γειτονία στην νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ανατολική περιοχή και την ανατολική γειτονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την ερώτησή σας για μια διεθνή συμφωνία η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο αν θέλετε νομικό πλαίσιο το οποίο θα διαδεχθεί τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου και θα εξασφαλίσει και τα κατάλληλα κονδύλια και το προσωπικό. Αυτό λοιπόν το ζήτημα τέθηκε ε, μεταξύ των μελών ε, του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά δεν έχει επιτευχθεί μια ομοφωνία γιατί πρόκειται βέβαια για μια χρονοβόρα διαδικασία αλλά και πολιτικά ευαίσθητη. Οπότε παρότι θα μπορούσε να αποτελέσει μακροπρόθεσμα τουλάχιστον ε, αυτή η λύση μια βιώσιμη εναλλακτική αυτή τη στιγμή δεν, μπορεί, ε, δεν θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί. Όμως μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει λοιπόν την οικονομική βιωσιμότητα. Η ε, χρηματοδότηση των προγραμμάτων που σήμερα ε, υλοποιεί βασίζεται στη χρηματοδότηση των κρατομέλων και από εκεί και μετά η βιωσιμότητα σε επίπεδο προσωπικού βασίζεται σε περαιτέρω χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και ο κύριος Λάμστορφ, μια ε, ε, απόσπαση, ε, κάποιες αποσπάσεις γίνονται ενίοτε από την πλευρά των κρατών μελών όπως αναφέρθηκε δηλαδή πρόσφατα από τη Δανία. Ε, υπήρξε απόσπαση ενός ειδικού. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, τις δικές μας, τα δικά μας σχόλια σε ό,τι αφορά ε, την προπαγάνδα ή την ε, έλλειψη ισορροπία σε ό,τι αφορά την ενημέρωση από πλευρά των μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας. Ναι, εγώ θεωρώ πως η ορολογία που ζητούμε, που, χρησιμοποιούμε εδώ θα, είναι η ενδεδειγμένη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το Ισλαμικό κράτος και τα σχετικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ε, ε, για παράδειγμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ε, στην Ρωσία έχουμε μια προπαγάνδα κρατική αν θέλουμε ενώ από την πλευρά του Ισλαμικού κράτους έχουμε μια προπαγάνδα που προέρχεται από έναν τύπο, από ένα τύπο σέκτας η οποία προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους οπαδούς. Από πλευρά λοιπόν μεθοδολογία, δεν θεωρούμε πω αυτά τα δύο είδη προπαγάνδα αποτελούν το ίδιο και το αυτό και κατά συνέπεια διαφορετικέ μεθοδολογίε θα πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση, για την καταπολέμησή του. Πάντω, σίγουρα χρειαζόμαστε μια οριστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία μα. Τώρα ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πανσέρη ε, για τα θετικά του σχόλια και για τι ε, καλέ ειδήσει που ακούσαμε, δηλαδή ότι θα εξετάσει ε, μια ε, ε, υποστήριξη του Ταμείου από την πλευρά της. Ε, μου θέσατε ένα ερώτημα ως προς το πού θα πρέπει να επενδύσουμε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες μας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την νότια κοιτωνία Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε ήδη στο 2016, δηλαδή η έκθεση αναφέρεται στο 2015, αλλά δεν μπορούμε βέβαια να την αποσπάσουμε από τόσα συνεχίζουν να συμβαίνουν σήμερα μέσα στο 2016. Οπότε λοιπόν εγώ θεωρώ πως οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία, στο Λίβανο και αλλού θα πρέπει να αναφέρονται και θα πρέπει να ε, κάνουμε και περισσότερα project, να κάνουμε περισσότερες δράσεις, γιατί πραγματικά δεν το έχουμε κάνει ε, επαρκώς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να εστιάσουμε στην ανθρωπιστική ε, πτυχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να κερδίσουμε αν θέλετε ε, και την εύνοια, την συμπάθεια των ανθρώπων η οποία δηλαδή όλο ένα και περισσότερο ε, είναι πιο απογοητευμένοι συνεχίζουν να κατοικούν, να, να παραμένουν σε αυτούς τους καταπλησμούς τους ε, προσφυγικούς όπου ακόμα και η κάλυψη των βασικών τους αναγκών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όταν λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση εμείς δεν αξιοποιούμε την ευκαιρία για να προβληθούμε περισσότερο σε αυτά, σε αυτά τα σημεία του κόσμου ενδεχομένως να δημιουργήσουμε μια κατάσταση η οποία διατηρηθεί για μία σειρά ε, ετών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε εδώ στην νεολαία, στην ε, εκπαίδευση, στη μόρφωση των ανθρώπων οι οποίοι ελπίζουμε θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στη Συρία και οι οποία θα είναι, θα είναι αρμόδιοι για την ανοικοδόμηση εκ νέου αυτού του κράτους. Είναι μια χαμένη ευκαιρία να μην το κάνουμε λοιπόν και θα πρέπει να, το, να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Δεν λέω δηλαδή ότι δεν κάνουμε τίποτα τη σημερινή ημέρα, αλλά σας λέω ότι θα πρέπει περισσότερα προγράμματα, προγράμματα θα πρέπει να ξεκινήσουν εδώ, περισσότερα κονδύλια θα πρέπει να επενδυθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ε, η Λιβύη αποτελεί και πάλι έναν τομέα τον έχουμε, ο οποίο καταλήψει ένα κράτο σε ό,τι για παράδειγμα την υποστήριξη τη μόρφωση, την υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών ε, και την ενίσχυση των μηχανισμών για την επίλυση των συγκρούσεων. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Αστροπίτσιους για, το, για την προοπτική που μας έθεσε, δηλαδή ε, το γεγονός ότι καλούμαστε να εργαστούμε σε μια ολοένα και δυσκολότερη χρονική συγκυρία. Δηλαδή ε, ε, το, τα περιθώρια αν θέλετε λοιπόν της κοινωνίας των πολιτών περιορίζονται ολοένα και περισσότερο και ε, τα όσα οι παράγονται από την ε, Ρωσία ε, συνεχίζουν να εξαπλώνονται και ε, σε μία σειρά από άλλες χώρες όπως το Αζερμπανιά και συνεχίζει να συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να το θέσουμε με σαφήνα. Η κοινωνία των πολιτών δεν αποτελεί απειλή για καμία κυβέρνηση. Οπότε θα πρέπει να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη δημιουργία τη κοινωνία των πολιτών, οπουδήποτε αυτή προσπαθεί να διαμορφωθεί. Και σε σχέση με αυτό το ερώτημα που τέθηκε σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των δικών μας, ε, αν θέλετε, αρχών, εμείς βασιζόμαστε πάντα σε αιτήματα. Δηλαδή μόνο αφού λάβουμε αίτημα εμείς ενεργοποιούμαστε με υποστήριξη και δεν ε, υποστηρίζουμε κάθε είδο δημοκρατία. Υποστηρίζουμε μόνο τι δημοκρατίες εκείνε οι οποίε υιοθετούν και ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες ε, που ακολουθούμε εμείς. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, τους τομείς όπου υπάρχει ιδιαίτερα εχθρικό περιβάλλον ε, και όταν λοιπόν μας ρωτάνε θα συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε ακόμα και αν το περιβάλλον γίνεται όλο και εχθρικότερο απέναντί σας εμείς τους λέμε ναι φυσικά θα συνεχίσουμε γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικό. Όταν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη από υποστήριξη και χρειάζονται υποστήριξη. Για παράδειγμα, και εγώ ε, ως ακτιβιστής κατά τη δεκαετία του 80 στην ε, Πολωνία, ε, προφανώς είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και υπήρχε βέβαια ο κίνδυνος να βρεθούμε φυλακισμένοι, οπότε όταν για παράδειγμα μου έστελνε κανείς ένα φωτοτυπικό ζήρουξ από την Δανία, ε, έκανε απλώς ε, και μόνο αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο, κάποια αρχή δημοκρατική την οποία εξήγαγε προς εμένα με αυτόν τον τρόπο. Ε, και αυτό ακριβώς ισχύει και για μας. Δηλαδή εμείς δεν λέμε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί συγκεκριμένα η προπαγάνδα της ουσίας. Υπάρχει υπήρχε μια συγκεκριμένη έκφραση που ακολουθούσαν τα μέσα ενημέρωσης και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας βασικός κεντρικός φορέας στη Ρωσία ε, στον τομέα της ενημέρωσης, πράγμα το οποίο βέβαια αντίκειται στην αρχή της πλουραλιστικότητας των μέσων ενημέρωσης. Και αυτό ακριβώς λέμε ότι ε, στη δική μας έκθεση ας μην καταπολεμούμε, ας μην γίνεται προσπάθεια καταπολέμησης της προπαγάνδας με αντιπροπαγάνδα. Δημιουργήστε λέμε περισσότερο, περισσότερα περιθώρια για να υπάρχει ακριβώς πλουραλισμός, να υπάρχουν περισσότεροι φορείς στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Άρα λοιπόν εκεί εμείς που προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε είναι η πρόσθεση των αξιών μας, όχι των συμφερόντων μας. Δεν μπορούμε εμείς να υποστηρίξουμε ούτως ή άλλως τα συμφέροντα κάποιου συγκεκριμένου κράτους μέλους, αν είναι, είτε είναι της Γερμανίας, ή της Ισπανίας ή οποιοδήποτε άλλο. Ουσιαστικά ε, έχουμε... Ε, κάποιες βασικές κοινέ αξίες τις οποίες προσπαθούμε να θεωρήσουμε και οι οποίες κοινέ για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να απάντησα σε όλα τα ερωτήματά σας και αν όχι με στη διάθεσή σας για να εξολογήσω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πομιανόφσκι που ήρθατε να μας παρουσιάσετε την ετήσια έκθεση και που καθίσατε και συζητήσατε μαζί μας. Θα περάσουμε στη συνέχεια στην συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο μετά από λίγα λεπτά. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt begrüßen. Ε, κύριε και κύριοι, σας καλωσορίζω για το επόμενο θέμα Έχουμε μαζί μας τον κύριο West Cote που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος τη Ευρωπαϊκής Περισσέως Εξωτερικής Δράσης για τη Βόρεια Αφρική και τον ε, κύριο ε, Κιόλα, ο οποίος είναι αρμόδιος για την νότια πολιτική γειτονία. Εδώ θα ασχοληθούμε βέβαια με την κατάσταση ε, τη σημερινή κατάσταση ε, στο Μαρόκο. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, ειδικότερα και μετά από την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικοστήριο σε ό,τι αφορά την υπόθεση που Ισάβιου κατά του Συμβουλίου και σε ποιο βαθμό δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια συμφωνία για τα ε, αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα της Αλίας και η περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Υπάρχει και η δυνατότητα βέβαια, εδώ θα υπάρξει η δυνατότητα ε, να ενημερωθούμε σχετικά με την επίσκεψη ε, ε, Πρόεδρου της Επιτροπής κυρίας Μογκερίνη στο Ραμπάτ στις 4 Μαρτίου και όπου βέβαια ακριβώς συζητήθηκε και αυτή η συμφωνία που μόλις ανέφερα. Το Μαρόκο λοιπόν έλαβε κάποιες αποφάσεις τις οποίες μας τις κοινοποίησε για διαστόματος ε, του Υπουργού Πολιτισμού. Ο Βασιλεύς Μοχάμεντ συγκάλεσε μια συνεδρία με τους υπουργούς ε, και τους ε, πρέσβες 6 Μαρτίου και με συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και ο κύριος Μπορίτα τώρα θα μας επισκεφθεί στα τέλη του μηνός Μαρτίου, μέσα στις επόμενες δηλαδή ημέρες, σε συνέχεια και εκείνη της ε, συνάντησης και θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν από πλευρά σας ε, τι θέλετε να κάνουμε από εδώ και στο εξή και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε δηλαδή στο Μαρόκο ότι ένα κράτο δικαίου δικαίου είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με αποφάσεις ενός δικαστηρίου χωρίς αυτό ε, χωρίς ε, υποχρεωτικά αυτή η απόφαση του δικαστηρίου να συμφωνεί με τα συμφέροντά του. Ότι δηλαδή είναι υποχρεωμένο να ε, συμμορφώνονται με τέτοιου είδου αποφάσεις είτε αυτή η απόφαση είναι υπέρ είτε κατά των συμφερόντων του λογοκράτους. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Westcourt. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαράξη να βρίσκομαι εδώ πέρα στην Επιτροπή σας. Ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που απευθύνω όμως στην Επιτροπή σας στο νέο μου ρόλο. Διευθύνων Σύμβουλος δηλαδή για την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εκ νέου στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας πω πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την κατάσταση των σχέσεών μας με το Μαρόκο. Το Μαρόκο, όπως το γνωρίζετε περισσότεροι, είναι ένας από τους πιο στενούς εταίρους που έχουμε στην περιοχή αυτή. Έχουμε πολύ ε, θετικές σχέσεις που καλύπτουν πολλούς τομείς. Έχουμε προφανώς την Συμφωνία Σύνδεσης, μια ευρύτατη εταιρική ε, συμφωνία που καλύπτει πάρα πολλούς τομείς, τομείς στους οποίους συνεργαζόμαστε στενά με το Μαρόκο και υπάρχουν και συγκεκριμένες επιτροπές συζήτησης. Καλύπτουμε το εμπόριο, τη γεωργία, την εμπορική δραστηριότητα, τον πολιτισμό, την καταπολέμηση τρομοκρατία, τη μετανάστευση, την ενέργεια και το καθεξής. Συνεργαζόμαστε λοιπόν πολύ στενά με το Μαρόκο σε πάρα πολλού τομεί και η συνεργασία αυτή πραγματικά ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και για τι δύο πλευρέ του παρελθόν. Τώρα, πώς έχει η σημερινή κατάσταση. Προέκυψε από μία απόφαση που έλαβε το Γενικό Δικαστήριο, το πρώην πρωτοδικείο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 10 Δεκεμβρίου. Απόφαση που έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου που εφαρμόζει την Αγροτική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Αποφάσισε λοιπόν το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει εν μέρη την συμφωνία αυτή και ιδίω το τμήμα εκείνο τη συμφωνία που έχει να κάνει με τη Δυτική Σαχάρα. Δεν θα περάσω στι λεπτομέρειε τη δικαστική αυτή απόφαση. Είναι δημόσιο το έγγραφο, μπορείτε να το συμβουλευτείτε εφόσον θέλετε. Προβλέπετε εκεί πέρα όλη η αιτιολόγηση του δικαστηρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το δικαστήριο είπε ότι ισχύει στο σύνολό τη η αγροτική αυτή συμφωνία. Υπάρχει πρόβλημα απλώ με το τμήμα εκείνο που είχε να κάνει με την Δυτική Σαχάρα. Αυτό θέτουν ένα αμφιβόλο και αυτό επιθυμεί να ακυρώσει το Γενικό Δικαστήριο. Είπα ότι εκπρόσωπο η κυρία Μογκερίνη έκανε ευθύ αμέσω μετά την απόφαση αυτή μια δήλωση, συζήτησε στη συνέχεια με τα κράτη-μέλη και στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι δεν συμφωνούμε με τη δικαστική αυτή απόφαση και ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να κάνουμε έφεση. Την απόφαση αυτή έλαβε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Δεκεμβρίου. Και είχαμε επίσης και συνεδρίαση του Συμβουλίου ε, Σύνδεσης, όπου συζητήθηκε το ζήτημα αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης που έχουμε προφανώς μαζί με το Μαρόκο, και είπαμε και εμεί τότε επίσημα προ το Μαρόκο ότι θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή του δικαστηρίου δεν πρόκειται να επηρεάσει την μακροχρόνια αυτή πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με τη χώρα αυτή. Είπαμε επίση ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι οι νομικέ συμφωνίε εξακολουθούν να ισχύουν και προφανώ πρέπει να συνεχιστεί και η συνεργασία. Στη συνέχεια Γίνανε πολλές έντονες συζητήσεις με την μαροκινή πλευρά, η οποία όπως καταλαβαίνετε είχε πάρα πολλά ερωτήματα πλέον σε σχέση με τη δικαστική αυτή απόφαση, σε σχέση με τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση αυτή από νομικής και πολιτικής πλευράς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των συζητήσεων αυτών εγώ πήγα στο Ραμπάτ, όπου γίνανε εκτενέστατες πολύ ωραίες συζητήσεις τον Δεκέμβριο του 2015 και έπειτα τον Φεβρουάριο να συμπορείτε, ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε, του Μαρόκου ήρθε στι Βρυξέλλε προκειμένου να αποσαφινιστούν περαιτέρω, περαιτέρω οι επιπτώσει τη δικαστική αυτή απόφαση. Όλα αυτά οδήγησαν στην επίσημη υποβολή της έφεσή μας από τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου κατά της δικαστικής αυτής απόφασης. Αυτό έγινε στις 19 Φεβρουαρίου και έπειτα στις 25 Φεβρουαρίου το Μαρόκο ανακοίνωσε ότι θεωρούσαν το ζήτημα αυτό ήταν τόσο σημαντικό για αυτούς που θα επιθυμούσαν τελικά να τονίσουν την σημασία της απόφασης αυτής παγώνοντας τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ζητήματα πέρα από τη δικαστική αυτή συμφωνία. Με την εξαίρεση μάλλον με συγχωρείτε της δικαστικής αυτής συμφωνίας. Έπειτα, μετά από συνεχιζόμενες επαφές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές, αποφασίσαμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος θα πήγαινε στο Ραμπάτα και ότι ο κύριος Μπουρίτα από την πλευρά του Μαρόκου θα ερχόταν στις Βρυξέλλες. Η πρώτη αυτή επίσκεψη έλαβε χώρα στις 4 Μαρτίου. Όντως η ύπατη εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μογκερίνη πήγε στο Ραμπάτ και είχε και εκεί εκτενείς επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου, τον κύριο Μεζουάρα και δώσανε στη συνέχεια κοινή συνέντευξη τύπου, στα πλαίσια τη οποία η κυρία Μογκερίνη είπε ότι η εταιρική σχέση που έχουμε με το Μαρόκο είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαίωσε επίση ότι εμεί θεωρούμε ότι η φυστάμενη συμφωνία εξακολουθεί και ισχύει από νομική πλευρά. Έχει επομένω μία, αποτελεί λοιπόν μία πολύ σημαντική βάση για την περαιτέρω συνεργασία μα με το Μαρόκο. Και είπε επίση η κυρία Μογκερίνη ότι θα αποκαταστήσουμε τις πλήρεις επαφές μας με το Μαρόκο και την πλήρη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, προκειμένου να δούμε τι μορφή θα πάρει η μελλοντική μας συνεργασία. Και προς τα τέλη του μήνα ο κύριος Μπουρίτα, ο Υπουργός Μπουρίτα θα έρθει στις Βρυξέλλες, προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που ξεκίνησε στι αρχέ Μαρτίου με την κυρία Μογκερίνη και προκειμένου να δούμε πώ θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε περαιτέρω λεπτομέρειε τη συνεργασία μα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την πλήρη συνεργασία μας με το Μαρόκο. Αυτή είναι η βασική επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Όπως σας είπα, αποκαταστήσαμε τις επαφές μας με το Μαρόκο. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τώρα πλήρως και τη συνεργασία μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να επιλύσουμε την νομική αυτή κατάσταση που έχει προκύψει το συντομότερο δυνατό. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα γίνει μέσω της επίσημης έφεσης που έχουμε υποβάλει προς το Γενικό Δικαστήριο. Αυτά κύριε Πρόεδρε, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και προφανώ είμαι στη διάθεση του συναδέλφου σα για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσει. Με την άδειά σα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μου κύριο Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, κύριε, θα κάνω κάποια συμπληρωματικά σχόλια στα όσα είπε ο συνάδελφος Νικόλα ω προ την οικονομική συνεργασία και χρηματοοικονομική συνεργασία με το Μαρόκο. Θα ξεκινήσω όμως λέγοντας ότι ε, ειδικότερα πέρυσι το 2015 η συνεργασία με το Μαρόκο ήταν πραγματικά υποδειγματική. Ε, το Μαρόκο έχει ε, ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση, επισήμως δηλαδή την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε ό,τι αφορά μια πλήρη και εμβαθυμένη συμφωνία ελευθέρω εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρότι δεν έγιναν επί της αρχής διαπραγματεύσεις ε, πέρυσι. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη χώρα της ευρύτερης περιοχής η οποία ξεκίνησε επισήμως αυτή τη διαδικασία. Επίσης ε, το 2015 όταν είχαμε, ε, συμβουλευθήκαμε στο πλαίσιο της Ανατολικής και Νότιας γειτονίας με τις διάφορες χώρες σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της ε, πολιτικής ε, γειτονίας, ε, το Μαρόκο πραγματικά συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση και υπήρξε ένα πολύ φιλόδοξο έγγραφο από την πλευρά του, το οποίο κατεδείκνει ότι αποφάσισε να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύνδεση προφανώς όχι ως κράτος μέλος, αλλά ε, μια σύνδεση, ε, αυξημένη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυγχρονισμού του, του, του, του, του Μαρόκου και πραγματικά αυτή η φιλοδοξία, αυτή η στάση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια προχωρημένη σχέση συνεργασίας και εμπορικής συνεργασίας με το Μαρόκο σε σύγκριση με άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά την ίδια τώρα τη συνεργασία, ε, ε, το 2015 μας οδήγησε σε νέα, νέους αριθμούς. Για παράδειγμα, το 2015 υπό το χρηματοδοτικό μέσο της ε, πολιτικής γειτονίας, το οποίο δεν είναι και το μόνο χρηματοδοτικό μέσο, 225 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για ε, χρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης, ε, ε, μεταρρύθμισης του σοφρονιστικού συστήματος, διακυβέρνησης και δικαιοσύνης, αλλά και στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών. Και αυτό οδήγησε σε καταβολή πληρωμών ε, της τάξης των 180 ε, με 190 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε αυτό ε, τι μας δείχνει ότι υπάρχει πραγματικά μια εντατική συνεργασία και μια θετική και επικοδομητική συνεργασία μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά εδώ έχει αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο το Μαρόκο στο πλαίσιο δηλαδή της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας. Τώρα με βάση τα όσα έλαβαν χώρα και τα οποία ε, ε, ε, στι τις τελευταίες εβδομάδες και σας τα εξήγησε ο συνάδελφος Μπέσκοφ μόλις τώρα, έχουμε βρεθεί σε μια κάπως δυσκολότερη θέση γιατί η άμεση αντίδραση ήταν ότι ε, η πλευρά του Μαρόκου αποφάσισε να παγώσει τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια σειρά εβδομάδων μετά από την επίσκεψη της Αντιπροέδρου και υψηλής εκπροσώπου ε, για τα ζητήματα της ε, εξωτερικής πολιτικής Μογερίνη στο Μαρόκο και μετά από την επίσκεψη του Υπουργού Μπορίτας στις Βρυξέλλες έχουμε μια προσπάθεια για να διευκρινιστεί λίγο η κατάσταση ως το που βρισκόμαστε και προκειμένου ακριβώς να ξεπαγώσουν αν θέλετε οι επαφές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, ε, η ε, εφαρμογή για αυτής της απόφασης ε, βέβαια από την πλευρά του Μαρόκου δεν έχει γίνει ομοιόμορφα από την πλευρά όλων των Υπουργείων. Δηλαδή και κατέστησε σαφές από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών τελευταία εβδομάδα δεν είναι και το ίδιο πεπισμένο ότι όλα τα Υπουργεία ακολουθούν αυτή την απόφαση η οποία λήφθηκε ω προ δηλαδή τι επαφέ και σε ποιο βαθμό αυτέ θα πρέπει να γίνονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να καταστήσω σαφέ εδώ στην αίθουσα είναι ότι εμεί δεν σταματήσαμε τη συνεργασία μα ούτε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το Μαρόκο από την πλευρά του. Όλοι μα δηλαδή ε, θέλουμε να συνεχιστεί η συνεργασία που έχουμε αλλά υπάρχουν προβλήματα γιατί σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν θέλουν να υπάρξει ιδιαίτερη προβολή των επαφών που λαμβάνουν χώρα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου και αυτό βέβαια αποτελεί και πηγή ε, παρανοήσεων τι οποίε ε, καλούμαστε να διευκρινίσουμε με την πλευρά του Μαρόκου. Για παράδειγμα, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να έχουμε τεχνικές, ε, τεχνική συνεργασία, δηλαδή συμβούλου οι οποίοι θα μπορούν να συναντούν του ομολόγου του στο Μαρόκο, τεχνικοί εμπειρογνώμονε οι οποίοι μπορούν να έχουν επαφή μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων όλα αυτά είναι σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν τόσο ώστε να συνεχιστεί και η ατζέντα της συνεργασία μας ε, και μέσα στο 2016. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν και αυτοί οι κίνδυνοι, ο ε, επικεφαλής ε, της δική μας αντισυκοσοπίας στις 12 Φεβρουαρίου απέστειλε μια ε, ε, επιστολή ε, στον Γενικό Διευθυντή του για ζητήματα οικονομικών της πλευράς του Μαρόκου, ο οποίος είναι αρμόδιος για, όλα τα, για όλες τις επαφές του Μαρόκου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπάθησε λοιπόν σε αυτή την επιστολή να εξηγήσει ποια είναι τα, οι περιορισμοί στο χρονοδιάγραμμά μας που μπορούν να προκύψουν εάν δεν συνεχίσουν οι τεχνικές διαβουλεύσεις στους διάφορους τομείς. Γνωρίζετε δηλαδή καλύτερα Όλοι σας από μένα ότι βασιζόμαστε επί τη βάση αιτήσεων προϋπολογισμών, δηλαδή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβλέπουν έναν προϋπολογισμό ε, για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία σε αιτήσια βάση ε, ε, προς την Επιτροπή και οτιδήποτε δηλαδή δεν αξιοποιηθεί ε, στο επίπεδο των μέσων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ουσιαστικά χάνεται, δηλαδή πέφτει θύμα αυτής της αιτήσιας οργάνωσης του προπολογισμού. Οπότε λοιπόν κάθε χρόνο είναι δύσκολο να ξεκινάμε να αναδιατυπώνουμε αν θέλετε το επίπεδο της εργασίας μας στο πλαίσιο για παράδειγμα νέων προγραμμάτων πλήρως τήρηση των σχετικών κριτηρίων και ούτω καθεξής. Ε, όσο λοιπόν ε, δεν προχωράμε φέτος, τόσο πιο σφιχτό θα είναι και το χρονοδιάγραμμά μας για την εφαρμογή των προγραμμάτων, τόσο λοιπόν πιο σφιχτά τα ε, περιθώρια για την αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων του, της, του χρηματοδοτικού μέσου της πολιτικής γειτονίας. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητήσαμε, τα αναφέραμε και στην επιστολή και 551 εκατομμύρια ευρώ αναφέραμε στο Μαρόκο ως σορευτικό ε, ως σωρευτικές δεσμεύσεις, αθρηστικές δεσμεύσεις για ε, προγράμματα και ε, δεσμεύσεις δηλαδή από πέρσι για προγράμματα τα οποία θα πρέπει να υπογραφούν αλλά και περαιτέρω προγράμματα που ξεκινούν φέτος για παράδειγμα σε ό,τι αφορά χρηματοδότηση προγραμμάτων υποδομών με χρηματοδότηση από πλευρά χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν και κάποιες δράσεις ε, οι οποίες έχουν ξεκινήσει και οι οποίες, ε, τις μας έχει πει το Μαρόκο πώς το ενδιαφέρον και πώς θα ήθελε να ε, συνεχιστούν ε, ταχύτατα. Και εδώ αναφερόμαστε στο twinning μεταξύ υπηρεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηρεσιών του Μαρόκου κάτι ακόμα που μπορεί να ενδιαφέρει ε, κάποιους ε, συναδέλφους ιδιαίτερα είναι ε, το διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ Ισπανίας, Πορτογαλίας και Μαρόκου και το οποίο θα πρέπει να και για το οποίο δηλαδή ε, πριν από τα τέλη του Μαρτίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικέ δεσμεύσει των κονδυλίων ε, του υπροπολογισμού για να μπορέσει να τρέξει. Άρα λοιπόν η πλευρά του Μαρόκου γνωρίζει καλά του περιορισμού που έχουμε σε επίπεδο χρονοδιαγράμματο για την εκτέλεση του υπροπολογισμού και ότι δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο από την πλευρά μα εμεί δεν, δεν παίζουμε παιχνίδια με την πλευρά του Μαρόκου. Δηλαδή είναι περιορισμοί αυτοί που υπάρχουν, είναι κατοχυρωμένε στι δικέ μα ε, συνθήκε στην, ε, στην εκτέλεση του προπολογισμού μα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε όσο πιο εντατικά γίνεται τις προσπάθειες ε, που έχουμε ξεκινήσει και μετά από την επίσκεψη της κυρία Μολιερίνης στο Ραβάτου, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών μα, όπως τις είχαμε προγραμματίσει και έτσι να ε, υπάρξουν και ε, τα, τα κατάλληλα κονδύλια τόσο ανάληψης υποχρεώσεων όσο και πληρωμών που θα εκτελεστούν στο σύνολό τους και σε υψηλότερο βαθμό από το 2015. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Εμείς είμαστε πολύ ε, φιλόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε στο, στους κανονικούς ρυθμούς της συνεργασίας μας, ώστε να καταστεί αυτό δυνατό. Σας ευχαριστώ. Κύριος Παντσέρη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν τρέφω καμία αμφιβολία για το ότι ε, όντω είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Και για μας δηλαδή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι είναι ένας προνομιακός στρατηγικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντως στο πλαίσιο της νέας κατάστασης που προέκυψε μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου που δεν αναγνωρίζει ένα τμήμα της Αγροτικής Συμφωνίας, ιδίως αυτό που έχει να κάνει με την Δυτική Σαχάρα, πρέπει να δούμε αν και εμεί φέρουμε κάποια ευθύνη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αν δεν επαληθεύσαμε σωστά τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν φέρουμε κι εμείς ένα μερίδιο της ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια της συζήτησης αυτής ανοίγονται δύο βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν ιδίω παρουσία του κ. Westcott και υπό το φως της επίσκεψης της ΥΠΑ εκπροσώπου στο Ραμπάτ, κίνηση που θεώρησε όταν ιδιαίτερα θετική. Όπως υπόθηκε, η μαροκινή κυβέρνηση μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου αποφάσισε να παγώσει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι από ό,τι φαίνεται μετά την επίσκεψη Μογκερίνη τα πράγματα κάπως έχουν βελτιωθεί. Επίσης, νομίζω ότι δεν θα ακολουθήσουν εύκολοι μήνες στο άμεσο μέλλον, καθότι έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο στο Μαρόκο και ξέρετε ότι εν γέννη οι εκλογές δεν βοηθούν πάρα πολύ στο να υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στο ποιος είναι φιλοευρωπαίος και λιγότερο φιλευρωπαίος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχουμε κι εμείς μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στους εταίρους μας στο, Μα... στο Μαρόκο, όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Προσπαθούμε κι εμείς να εξηγήσουμε στο Μαρόκο ότι ε, η δικαστική αρμοδιότητα, οι δικαστικοί θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν απόλυτα αυτόνομα και ανεξάρτητα, επομένω μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητε αποφάσει όπω αυτή η οποία λήφθη. Από την άλλη υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία θίξατε και εσεί και έχουν να κάνουν με το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, οι ερωτήσει μου έχουν να κάνουν με τα εξή σημεία. Πρώτον, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος που μπορεί να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση βάσει του ψηφίσματος 1754 των Ηνωμένων Εθνών. και δεν νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή η στάση που κράτησε το Μαρόκο απέναντι στον Πανκιμούν και δεν νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση. Όσο περνάει ο καιρός και όσο δεν διευθετείται το ζήτημα με τη Δυτική Σαχάρα, τόσο δυσχεραίνεται και εξέβρεση λύσης. Δεύτερον τώρα, εν αναμονή της επίλυσης σε όλα αυτά τα ζητήματα, εμείς δεν μπορούμε να παραπέουμε προς τη μία ή την άλλο πλευρά, θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή πολιτική στάση, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της περιφερειοποίησης ενέκρινε τη συμφωνία αυτή το Μαρόκο, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά ιδίω όσον αφορά το νότιο Μαρόκο ή τη Δυτική Σαχάρα, όπως θέλετε πείτε το, θα πρέπει να έχουμε μία κάποια αντιπαράθεση πλέον με την μαροκινή πλευρά, προκειμένου να έχουμε τουλάχιστον κάποιους θύλακες αυτονομίας στην περιοχή αυτή, όπως έχει γίνει πολλές φορές και με άλλες περιπτώσεις και με άλλες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι Ακόμα και στην αιτιολόγηση της δικαστικής απόφασης τίθεται το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, η έφεση που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή εμποδίζει και την Ελληνική Συμφωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε μία πολιτική αντιπαράθεση, ανταλλαγή απόψεων με τη μαροκινή πλευρά προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν και οι δύο συμφωνίες, και η Αγροτική και η ελληνική Συμφωνία. Ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχουν συμβάλει στο να καθυστερήσει η εξέβρεση λύσης. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η δική σας πρόταση σε σχέση με αυτά τα δύο δικά μου ερωτήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει η κυρία Γκάμπριελ. Θέλω να ευχαριστήσω και σας και την τη εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη για όλες τις προσπάθειες που έκανε να κρατήσει ως σημαντικό εταίρο το Μαρόκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι πολιτικά δεν μπορούμε να αφήσουμε το τελευταίο στάδιο της απόφασης να πλήξει τις μακρόχρονες σχέσεις μας με το Μαρόκο. Ένα κεφάλαιο που έχουμε χτίσει και δεν πρέπει να το καταστρέψουμε περιμένοντας την τελική απόφαση. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση τώρα επί της διαδικασίας. Σε τι βαθμό η διαδικασία που θα ακολουθήσει που είναι επιταχυμένη, είναι, κανονική, εξαρτάται και ο κάθε μήνας μετράει για μια εταιρική σχέση. Έπειτα, επιβεβαιώνω αυτά που είπε και ο κύριος Βέστκοκ, ότι το Μαρόκο είναι από τους πιο σημαντικούς και πιο σταθερούς μας εταίρους στην περιοχή. Γι' αυτό και έχουμε τομείς συνεργασίας που δεν πρέπει να πληγούν από την απόφαση αυτή. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ζωσπαστικοποίησης, ε, η σταθερότητα στην περιοχή, στην Αφρική εξαρτώνται από το Μαρόκο και ας μην ξεχνάμε και όσα έχει κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια για τη μετανάστευση το Μαρόκο και για την ασφάλεια. Σήμερα λοιπόν θέλω να με βεβαιώσετε ότι οι χώρες μέλη θα παραμείνουν ενωμένε. Είναι πολύ σημαντικό να μην ε, διχαστούμε πάνω σε αυτή την υπόθεση. Ήμασταν ε, σύμφωνοι όλοι στην αρχή και ελπίζω να παραμείνουμε έτσι. Έπειτα αυτή την κρίση μπορούμε να τη δούμε και σαν εφαλτήριο για να προχωρήσουμε περισσότερο, να ενισχύσουμε το πολιτικό διάλογο και να επικεντρωθούμε ε, στο θέμα του πώς θα προλαβαίνουμε τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν καλός συντονισμός και με τα μηνύματα που έρχονται από άλλα θεσμικά όργανα, από τα Ηνωμένα Έθνη, για παράδειγμα. Και ένα άλλο ζήτημα Ακόμα και αν σύμφωνα με τον Ευρωπαίο νομοθέτη η συμφωνία συνάδει με το διεθνές δίκαιο, όπως υπενθύμησε η κυρία Μακεβίνη στο Ραμπάτ, τι θα κάνει η Επιτροπή και το Συμβούλιο αν ε, στο εφετείο επιβεβαιωθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τι θα κάνουμε για να μην αμφισβητηθούν άλλες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο και πώς θα προσαρμοστεί η συμφωνία αυτή για να διασφαλιστούν τα ομοιβαία ωφέλη. Όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα, η απόφαση του δικαστηριού παραδόξως μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα, την απογραφή του πληθυσμού στο καταβλισμό Καλούφ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δούμε που πάει ανθρωπιστική βοήθεια επίσης. Ε, και τρίτον, να φροντίσουμε να τηρούνται τα ψηφίσματα των ΟΕΕ επικοδομητικά και αμερόληπτα. Επικοδομητικά και αμερόληπτα. Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη διαδικασία. Το κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μην μας επηρεάσουν ε, πράγματα αρνητικά στη διαδικασία αυτή και πάψουμε να είμαστε αμερόληπτοι. Ο κύριος Κούς, ευχαριστώ πρόεδρε. Για τη χώρα μου, ξέρετε, ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Σαχάρα είναι ευαίσθητο. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ειλικρινά με λυπεί να βλέπω πώς συμπεριφέρεται το Μαρόκο, σαν ένα κακομαθημένο παιδί. Άμα δεν του αρέσει μια δικαστική απόφαση, τα βάζει με μας. Ωραία. Είναι σημαντικός εταίρος, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, συμπεριφέρεται με σωστό τρόπο, τα δικαστήρια αποφασίζουν. Φυσικά πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους. Όμως το τελευταίο καιρό βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να δέχεται απαράδεκτες πολιτικές από κάποιες χώρες όπως είναι η Τουρκία και το Μαρόκο. Πρέπει να τα συζητάμε αυτά. Στο Μαρόκο πρέπει να εξηγήσουμε ότι στις σχέσεις μας πρέπει να κυριαρχεί ο σεβασμός και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά από τρία χρόνια φυλακή, οι φυλακισμένοι Σαραουί εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι για εβδομάδες. Πρέπει επίσης να πούμε στο Μαρόκο ότι πρέπει να σέβεται και την διεθνή νομιμότητα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπει να αντιβαίνει το Μαρόκο στην, ε, στα όσα λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για την, ε, από, τον αποεπικισμό της Δυτικής Σαχάρας. Η προσφυγή αυτή ομόφωνα γιατί. Πώς το βλέπει το Συμβούλιο και κάνει αυτή την προσφυγή. Έχουμε κάποιες αποφάσεις Λέμε ότι κάποιες είναι πολύ αυστηρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τι θα κάνει για αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή για να πάψει ο επικισμός στην περιοχή. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σουηδικά θα μιλήσω, αλλά βλέπω ότι φοράτε τα ακουστικά σας, οπότε εντάξει. Ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, Πολύ με ξέπληξε η απόφαση αυτή του είναι η ίδια ερμηνεία της σουηδικής κυβέρνησης, είτε αυτή είναι δεξιά είτε αριστερή. Για χρόνια υπάρχει κατοχή στη Δυτική Σαχάρα, το Μαρόκο είναι κατοχική δύναμη, δεν έχει λοιπόν το δικαίωμα να πουλάει ούτε να κάνει τίποτα με τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Και αυτό λοιπόν, αυτή η απόφαση δεν με εξέπληξε. Μάλιστα, χαίρομαι γιατί όντως μιλάει για την κατάσταση έτσι όπως ακριβώς έχει. Δεν μιλάει μόνο για τη συνεργασία με το Μαρόκο, αλλά γενικά όταν μιλάμε για το Μαρόκο δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τη Δυτική Σαχάρα. Είναι κατεχόμενα εδάφη και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Γιατί το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις η χώρα κατοχής στο Μαρόκο να μην έχει λόγο στα εδάφη αυτά. Και κάτι ακόμα, όλε οι χώρες, λέτε, συμφώνησαν. Δεν μπορώ να πω παρά για τη χώρα μου μόνο, όπου εμείς είχαμε διαφορετική άποψη για την συμφωνία, για τη Γεωργία, για την Αλία. Ακόμα και αν η Σουηδία συμφωνεί τελικά με αυτήν την δράση για να ξεμπλοκαριστεί η κατάσταση, δεν σημαίνει όμως ότι συγχρόνως συμφωνούμε με την γενική ερμηνεία. Όχι, πρέπει να δούμε τι γίνεται επί Καλό θα ήταν να υπάρχει μια ανώτερη, ανώτερη αρχή. Ω Σουηδία, πάντως, θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη μας τα όσα λέει και ο πληθυσμός επιτόπου. Υπάρχει απόφαση και από εκεί και πέρα να δούμε τι λένε οι πολιτικοί. Κάποιοι λένε ότι είναι κακομαθημένο παιδί το Μαρόκο, μπορεί. Εμείς πάντως το διεθνές δίκαιο πρέπει να υποστηρίξουμε και τη δικιά μας την εκτίμηση. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Τι γίνεται με την εφαρμογή της δικαστικής αυτής απόφασης. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Τώρα όμως ποια είναι ακριβώς η κατάσταση. Έχουμε προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και φτάνουν στην Ευρώπη και φέρουν ετικέτα, στην ετικέτα προέλευση Μαρόκο. Δεν θα ήταν σωστό αυτό. Δεύτερον, αυτά που διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωση του Μαρόκο, ο κυρία Μογκερίνη λέει ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο να συνεργαστούν για την ε, έφεση αυτή. Μα έτσι είναι σαν να νομιμοποιούμε μια κατοχική δύναμη και τη δράση της. Εντάξει, να συνεργαζόμαστε με το Μαρόκο για να λυθεί το θέμα της έφεσης, αλλά όχι έτσι συνεργασία. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο, με διακόπτει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι από την πλευρά μου, αλλά περιμένει και ο Επίτροπος έξω, οπότε θα πρέπει πραγματικά να περιορίσουμε το χρόνο αγόρευσης. Οπότε, κύριε Χάουιτ, είστε ο επόμενος στο κατάλογο των ομιλητών μου. Μπορείτε να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση, αλλά να μην μιλάμε μόνο για τη δικαστική απόφαση, να μιλάμε για τις σχέσεις μας με το Μαρόκο, την στρατηγική για τη δημοκρατία, ε, τη στήριξη της χώρας κτλ. Στη συζήτηση παγιδευόμαστε μερικές φορές και δεν συμφωνώ με όσα είπαν συνάδελφοι πριν. Πρέπει να δούμε τι είδους σχέσεις θέλουμε με το Μαρόκο. Αυτό είναι το βασικό. Και βρήκα ότι είναι πολύ σωστό αυτό που είπε η κυρία Μογκερίνη και η Κομισιόν όσον αφορά την έφεση, αλλά από την άλλη μεριά να φροντίσουμε οι δικές μας αρχές να τηρούνται. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να κρίνουν κάθε φορά αν τηρείται το διεθνές δίκαιο ή όχι, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μεροληπτούμε. Ούτε ο κύριος Βέσκοτ, ούτε ο κύριος Κούλερ είπε τι κάνουμε για την επίλυση της διένεξης όσον αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπανκιμούν ε, εξέφρασε επικρίσεις σε βάρος του Μαρόκου δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιφάσκει με τις θέσεις των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι είπε ο κ. Παντζέρη να πάει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Σαχάρα. Ναι, να γίνει. ο Αραβικός Σύνδεσμος επίσης ασχολείται με το θέμα και εμείς θέλουμε το Μαρόκο να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αραβικής λύσης. Άρα όταν τίθονται τέτοια ζητήματα εμείς θα τα υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. ένα λεπτό ο καθένας αλλιώς θα σταματήσω απλά την ε, συζήτηση και δεν θα συνεχίσουμε το κατάλογο των μιλητών. Ευχαριστώ τους ε, μιλητές μας για τόσο μας είπαν. Το ότι είπα κύριε Μογκερίνη στο μαράκι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση για το Μαρόκο, να μην υπάρχουν παρεξηγήσει και η επικοινωνία μεταξύ μας να είναι ομαλή. Το Μαρόκο είναι πολύ σημαντικός εταίρος, όπως είπαμε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της έχει μια, ένα προθυμένο καθεστώς ε, σύνδεσης, είναι τέρο στρατηγικής σημασίας, λέμε, το Μαρόκο, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα της μετανάστευσης, της ασφάλειας, καταπολέμησης, της τρομοκρατίας και πολλών άλλων, ε, οικονομία κλπ. κλπ. Και σίγουρα το Μαρόκο πρέπει να κάνει πολλά για το διεθνές δίκαιο, πρέπει να επαναλάβουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση μας μαζί του, που απορρέουν από πολλά χρόνια πριν κοινή δράση και η εμπειρία μας είναι θετική να μην περιοριζόμαστε σε συγκυριακές δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει έφεση, ομόφωνα μάλιστα, στην ε, δικαστική αυτή απόφαση. Η σχέση αυτή πρέπει να συνεχίσει σε θετική νότα, όπως μας παρουσίασαν και οι δύο μιλητέ μας και να μην επηρεαστούμε από τι δυσκολίε των τελευταίων ημερών. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, μόλις σας ανακοίνωσα ότι θα πρέπει να σταματήσουμε άμεσα τη συζήτησή μας, οπότε δεν θα μπορώ να επιτρέψω στους όλους τους ομιλητές από πάρουν τον λόγο. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκούρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πούμε ότι όντως το Μαρόκο είναι μία από τις πιο σταθερές χώρες της Βόρειας Αφρικής. Είναι πολύχρονος εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι επίσης και μία χώρα η οποία κάνει πολύ θετικές μεταρρυθμίσεις και αυτό πρέπει να το πούμε και επιφέρει πολύ σημαντικές ε, κοινωνικές αλλαγές επίσης. Για παράδειγμα, η θέση της γυναίκας στο Μαρόκο έχει αλλάξει πάρα πολύ με την πρόσφατη κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές που έχει κάνει η τελευταία κυβέρνηση και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε και τη χώρα αυτή και να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με αυτή τη χώρα. Και νομίζω ότι ε, η κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή αποτελεί δοκιμασία πραγματικά της συνεργασίας και της πολιτικής βούλησης της δικής μας. Μπορούμε τελικά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των εταίρων μας ή όχι. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, όλοι γνωρίζουμε πως έχουν τα πράγματα. Ξέρετε ότι στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στα πλαίσια της συνεργασίας με το Μαρόκο είχαν απόλυτη γνώση της κατάστασης στη Δυτική Σαχάρα και ποια είναι η τοποθέτηση του Μαρόκου σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Ενδεχομένω να δίστανται απόψει όσον αφορά την επίλυση τη διένεξη αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση αναφίβολα το Μαρόκο είναι η πιο σταθερή χώρα της Βόρειας Αφρικής και συμβάλλει πάρα πολύ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι επίσης μια χώρα η οποία ακολουθεί μια πολύ επικοδομητική πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης. Και έχουμε επίσης πάρα πολύ θετικές σχέσεις με το Μαρόκο σε σχέση με τους πρόσφυγες που έρχονται από το Μαρόκο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι επικοδομητική η σχέση που έχουμε με τη χώρα αυτή. Dankeschön, Herr Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι καταρχήν ε, ότι σας ζητώ συγγνώμη γιατί ήρθα τελευταία πιο άλλη σημαντική υποχρέωση. Απλώς θα ήθελα να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση κάνοντας μόνο ένα σχόλιο. Θα πρέπει να σεβαστούμε, θα πρέπει να γίνει σεβαστή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, γιατί είναι το δικό μας δικαστήριο της Ένωσης και κατά συνέπεια η Επιτροπή θα πρέπει να σεβαστεί αυτή την απόφαση. Οπότε ε, διαρωτώ με πώς η Επιτροπή τόσο γρήγορα ε, προέβη κατά κάποιο τρόπο σε μια αμφισβήτηση αν θέλετε αυτής της απόφασης ε, δηλαδή ε, προφανώς εμπόμαστε την σημασία του Μαρόκου αλλά και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κατους δικαίων είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα για μας και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας αποτελεί πραγματικά μια κραυγαλαία περίπτωση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κύριος Μποργέτζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό καταδεικνύει κατάφορα θεωρώ και νομίζω ότι το παραδέχονται αυτό και οι παρατηρητές από το ίδιο το Μαρόκο ότι ε, ο ρόλος του ε, δικαστηρίου αυτή τη στιγμή τίθεται να αμφιβόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά λειτουργήσε ως ένα παράλληλο κοινοβούλιο. Εμείς συντοποιείται ότι έχουμε συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προέρχονται και από πάρα πολλές αποφάσεις και από την ίδια την ομολογία του Γενικού Δικαστηρίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ότι αντί να κάνουμε εμείς εξωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική κάνει το Γενικό Δικαστήριο. Τι εικόνα δίνουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργώντα κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι γνωρίζαμε, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, ποια είναι η στάση διεθνής του Μαρόκο σε σχέση με την Δυτική Σαχάρα. Παρ' όλα αυτά υπογράψαμε καιροσκοπικά, με ιστοροβουλία θα έλεγα, μια συμφωνία, εθελοτυφλώντας για το πολιτικό αυτό ζήτημα το οποίο εκρεμεί. Αυτή τη στιγμή νομίζω πραγματικά όμως ότι η παρέμβαση της κυρίας Μογκερίνη έρχεται πάρα πολύ αργά και ουσιαστικά λάθος έχουμε κάνει εμείς. Εμείς θα έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη από το Μαρόκο για τη διεθνή αυτή γκάφα που κάναμε και την οποία προκαλέσαμε κιόλας. Ας μην ξεχνάμε ότι το Μαρόκο είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος, έχουμε όμως και πάρα πολλούς άλλους φίλους. Ας προσπαθήσουμε και το Μαρόκο και τους άλλους συνεργάτες μας στην καταπολέμηση τρομοκρατίας και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού να τους διατηρήσουμε. Merci Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να ακούγεται ότι το διεθνές δίκαιο είναι κατά του Μαρόκο στην υπόθεση αυτή που αφορά τη Σαχάρα. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συμφωνίες όλα αυτά τα χρόνια που δείχνει ότι το Μαρόκο διαθέτει νομικά επιχειρήματα για να αιτιολογήσει την κυριαρχία του στη Δυτική Σαχάρα. Και εγώ για χρόνια ε, πήγαινα στην τέταρτη, τέταρτη επιτροπή όσον αφορά τις απικίες του ΟΙΕ. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα και κατά τη διάρκεια της ιστορίας έχει επιχειρήματα μαζέψει το Μαρόκο για να πει ότι έχει κυριαρχία εκεί και ότι δεν πρόκειται για κατοχή. Άρα είναι επίμαχο το ζήτημα. Δεύτερον, το Μαρόκο αποτελεί έναν βασικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα σταθερό εταίρο, έναν εταίρο που έχει δείξει τις ικανότητες εκδημοκρατισμού που έχει, σεβασμού του κράτους δικαίου, καταπολέμησης τρομοκρατίας κτλ. και χρειαζόμαστε αυτό τον εταίρο στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ το μήνυμα της συμφωνίας αυτής δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικαθίσταται ουσιαστικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε θέματα ε, διεθνούς ε, πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και ότι τελικά μας αντικαθιστά. Καταλαβαίνω την αντίδραση του Μαρόκο. Μπορεί να φαίνεται κάπως απότομη, αλλά γιατί, γιατί θεώρησε ότι πρόκειται για προσβολή. Οπότε χαιρετίζω τις προσπάθειες της κυρίας Μογκερίνη για να διορθώσει την κατάσταση και καλώ τους συναδέρφους να καταλάβουν ότι επήγει η αποκατάσταση των σχέσεών μας με το Μαρόκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει και ο κύριος Πρέντα. Πρώτα απ' όλα, με εξέπληξε που είδα τις τελευταίες εξελίξεις με τον Πάνκι Μουν, ο οποίος μετά από ένα σοβαρό λάθος που έκανε, εξακολουθεί να επιδεικνύει νευρικότητα. Είπε στον, έδειξε μάλλον ότι εξακολουθεί να μην αισθάνεται άνετα στις επαφές του με τον Υπουργό Εξωτερικών, έκανε μια κάφα και είδαμε που οδήγησε σε τι αντιδράσεις. Είναι δυνατόν ο Γενικός ο Γραμματέας να χρησιμοποιεί τον όρο κατοχή. Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιεί αυτό τον όρο. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί μετά ξεπλάγει από την αντίδραση του Μαρόκου. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βουιστικότ να μας πει ποια είναι τα επόμενα στάδια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Σχέσης για τις σχέσεις μας με το Μαρόκο, χαιρετίζοντα βέβαια την χειρονομία της κυρίας Μογκερίνη που πήγε επί τόπου. Ο κύριος Παρνιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ναι, πολύ σύντομα τέσσερα θέματα θέλω να θίξω μαζί σας. Πρώτον, το ξέρουμε ότι η πολιτική εμπλοκή σε θέματα ασφάλειας του Μαρόκου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζουμε εμείς στη Γαλλία αυτό πάρα πολύ καλά, λαμβάνοντας υπόψη μας τι έγινε στη Γαλλία στις 13 Νοεμβρίου. Το πάγωμα λοιπόν διπλωματικών σχέσεων θα έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε τι μέτρα θα πάρετε προκειμένου το πάγωμα αυτό των σχέσεων να μην ζημιώσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ασφαλειά μας. Δεύτερον, είπατε πριν ότι το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του Μαρόκο. Όχι, εγώ νομίζω ότι βρίσκεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μπαλάκι. Εξάλλου το δικαστήριο στην απόφαση του το λέει λέει ότι πρόκειται για κάποιες ελλείψεις στα πλαίσια της Αγροτικής Συμφωνίας, ελλείψεις από πλευράς του Συμβουλίου. Οπότε, τι απαντήσεις θα δώσετε, τι θα κάνετε, ώστε να επωφελείται ο ντόπιο πληθυσμό. Τι θα κάνετε. Τρίτον, συνεργασία στο μεταναστευτικό. Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Είδαμε τα τελευταία χρόνια τι κατάφερε να κάνει το Μαρόκο. Είχαμε λοιπόν μεταναστευτική συνεργασία που στα γνωστά σημερινά πλαίσια είναι ουσιώδης. Οπότε τι προτείνεται στα πλαίσια αυτής της μεταναστευτικής συνεργασίας δεδομένου του παγώματος. Και όσον αφορά την επίλυση του, της διάνεξης για τη Δυτική Σαχάρα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι. Πρόκειται για πρόταση του Μαρόκου. Όπως εδώ και πολύ καιρό το έχει πει ο ΙΕ, πρόκειται για μια αξιόπιστη λύση. Μια προωθημένη αυτονομία δηλαδή στη Σαχάρα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν προτάσεις και από την ευρωπαϊκή διπλωματία, ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα πλέον να βγούμε από αυτά τα 40 χρόνια αδιέξοδο στο διπλωματικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθώς κανένας από σας δεν τήρησε το όριο του ενός λεπτού, θα πρέπει να διακόψω δυστυχώς αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Οπότε όσοι ε, δεν ε, θα πάρουν το λόγο και θα καταφέρουν να πάρουν το λόγο, ε, τους ζητώ να απευθυνθούν στους συναδέλφους από την ίδια πολιτική ομάδα που δεν τους επέτρεψαν. Να δώσω όμως τώρα το λόγο στον κύριο Westcott. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έκαναν τα σχόλιά τους και έθεσαν ερωτήματα. Πέντε σημεία θα ήθελα να θέσω, έτσι, απαντώντας τα όσα υπόθηκαν. Καταρχήν, να πω ότι αναγνωρίζω και εγώ πως ε, πολλοί από σας είπατε αποτελεί ένα στου πλέον στενού μα εταίρου στο πλαίσιο τη συνεργασία, και θα πρέπει να συζητούμε, ε, συζητήσουμε από κοινού κάποια ζητήματα που έχουμε. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ στενή συνεργασία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατία και θα πρέπει να την εμβαθύνουμε. Μετανάστευση είναι ένα δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλουμε να εμβαθύνουμε μια ήδη στενή συνεργασία που έχουμε αποτελεί δηλαδή ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για εμά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θέλουμε να έχουμε ένα πλήρε καθεστώ συνεργασία για τα ζητήματα τη μετανάστευση. Επειδή τώρα αυτή η σχέση μα ε, είναι σημαντική και για τι δύο πλευρέ, θα πρέπει και οι δύο λοιπόν, πλευρές, και το Μαρόκο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ε, συνεχίσουν να έχουν την κατάλληλη ε, εικόνα στο μέλλον ω προ το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ένα δεύτερο σχόλιο που θα πρέπει ε, θα ήθελα να κάνω είναι αυτό που αναφέρεται στο, στο, στο πρόβλημα της ε, Δυτικής ε, Σαχάρας και το οποίο αναφέρθηκε από πολλούς από εσά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αθετήσει εδώ και μία σειρά ετών μία πολύ σαφή στάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας. Και αυτή είναι ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες που κάνουν τα Ηνωμένα έθνη προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη και μακρόχρονη λύση η οποία θα προβλέπει την, τον αυτοπλουσιασμό των και την αυτοδιάθεση ε, του λαού της ε, Δυτικής ε, Σαχάρας με βάση και τις αρχές όπως αυτές έχουν κατοχυρωθεί και από την πλευρά των Ηνωμένων και θα προσπαθήσουμε όπως είπε και ο κύριος Γκάμπριελ από κοινού να επιτύχουμε μια λύση που θα κινείται σε αυτόν τον άξονα. Όπως ο Γάλλος συναδελφός πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο δεν θέλω να το υπεραπλουστεύσω εδώ αλλά είμαστε, βρισκόμαστε σε ε, στενές επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη και συναντήμαστε συχνά με τον Αναπλούδη Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Γραμματέα, οπότε υπάρχουν εδώ επαφές οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Ένα τρίτο ζήτημα τώρα είναι αυτό της νομικής διαδικασίας. Αντιλαμβάνομαι ότι η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ε, ζήτησε μια επιταχυμένη διαδικασία και αυτό γιατί τα, οι νομικές επιτυχίες εδώ είναι πολύ σημαντικές και είναι σημαντικό να επιληθούν το ταχύτερο δυνατό και αυτό ισχύει βέβαια και στο πλαίσιο ακριβώς της σχέσης μας με το Μαρόκο. Παρότι Παρ' αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η απόφαση ε, που εξέδωσε το δικαστήριο είναι κάπως περιορισμένη σε ό,τι αφορά το εύρος. Επειδή όμως δεν είμαι εγώ δεν θέλω να υπεραπλουστεύσω εδώ τα όσα αναφέρει η απόφαση, αλλά όπως ήδη υπόθηκε ουσιαστικά η απόφαση ε, ουσιαστικά λέει ότι δεν ε, μπορούν ε, να περιληφθεί αυτή η συγκεκριμένη περιοχή. Δεν αναφέρεται δηλαδή στο ότι δεν μπορούν να, να συμπεριληφθούν στην Συμφωνία Συνεργασίας με το Μαρόκο συγκεκριμένες περιοχές, απλά θα πρέπει να φροντίζουμε ότι ε, λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των λαών σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό ε, θέτει μια, ε, μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Ποιος μπορεί για παράδειγμα να κινηθεί νομικά εναντίον αυτής της απόφασης. Ποια, ποιο είναι το νομικό καθεστώς, αν θέλετε, τη νομική ισχύ τέτοιων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Αλλά αυτά βέβαια είναι πιο γενικά ζητήματα που τίθενται και προφανώς εμπειρογνώμονες σε αυτά τα νομικά ζητήματα μπορούν να το συζητήσουν περαιτέρω. Τέταρτο σημείο ε, το Μαρόκο δεν αποτελεί άμεσα συμβαλόμενο μέρος, αν θέλετε, σε αυτή τη συμφωνία. Ή μάλλον, συγγνώμη, στην, ε, στην ε, δικαστική υπόθεση, αλλά προφανώς έμεσα το ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και γι' αυτό έχουμε ακριβώς αυτόν τον εντατικό διάλογο με το Μαρόκο, ο οποίος συνεχίζεται. Γιατί δηλαδή το Μαρόκο θα πρέπει να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τι, τι ακριβώς συνιστά αυτή η απόφαση του δικαστηρίου. Και μας ενδιαφέρει και εμά. Και ως ένα καλό εταίρο δηλαδή, στο πλαίσιο τη συνεργασία μα. Θέλουμε να συνεχίσουμε ακριβώ τι επαφέ μα για να βοηθήσουμε το Μαρόκο να καταλάβει ποιο ε, θα μπορούσε να είναι δυνητικά ο αντίκτυπο αυτή τη απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προσφυγή και το ποια θα είναι η απόφαση που θα εκδώσει σχετικά το δικαστήριο, δεν γνωρίζω βέβαια, δεν έχω καμία ιδέα. Οπότε δεν θα προβώ σε περαιτέρω σχόλια σε σχέση με την απόφαση την ίδια και το ποιε είναι οι επιπτώσει αυτή τη απόφαση. Όμω, Προφανώ ισχύει το κράτο δικαίου και κατά συνέπεια σεβόμαστε τι αποφάσει που εκδίδει το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφώ, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αυτό και από εκεί και μετά να διευκρινιστεί δηλαδή το τι ακριβώ αναφέρει η απόφαση και από εκεί και μετά θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Και από εκεί και μετά βέβαια. Ε, ε, ε τι γίνεται στο επίπεδο τελικά τη συνεργασία μετά την απόφαση με το Μαρό. καταρχήν α επανέλθουμε εκεί που βρισκόμασταν. Στο επίπεδο δηλαδή τη συνεργασία ε, που είχαμε. Καταρχήν να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την ε, συνεργασία μας και θέλουμε από εκεί και μετά και να την εμπαθύνουμε όπως ήδη αναφέρθηκε και από τον ε, συναλφό λαό και από εσάς, από διάφορους αποβουλευτές. Υπάρχουν δηλαδή μια, ε, ένας αυξανόμενος αριθμός προβλημάτων τα οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού με το Μαρόκο. Θέλουμε να συνεχίσουμε για παράδειγμα τις τη της του, ώστε να συζητήσουμε και το, στο επίπεδο της αυξημένη κινητικότητα. αλλά βέβαια θα πρέπει να συνεργαστούν και οι δύο πλευρές για να επιτευχθεί εδώ κάποια πρόοδος. Οπότε με αυτό το σκεπτικό συνεχίζουμε. Εγώ πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Βέσκοτ ε, κάλυψε τα περισσότερα πράγματα. Στις ε, παρεμβάσεις σας ε, αναφερθήκατε στο ότι ε, η στρατηγική αυτή μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους δεν βρισκόμαστε στο κλασικό σενάριο της αναπτυξιακής βοήθειας. Έχουμε μία χρηματοδότηση κοινών δράσεων προς το κοινό συμφέρον. Ρωτήσατε τι πρόκειται να κάνουμε για τη μετανάστευση. Στα προγράμματα προβλέπουμε για το 2016 προβλέπεται να υποστηρίξουμε προγράμματα για την πολιτική μετανάστευση του Μαρόκου. 35 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια. Η συνεργασία λοιπόν αυτή είναι αμοιβαίως επωφελής. Και αυτό είναι και το κοινό μας συμφέρον. Θα πρέπει βέβαια συνεργασία να βασίζεται σε κοινή νομική κατανόηση των πραγμάτων. Ο Νίκ είπε ότι βάσει της νομικής αυτής απόφασης άλλωστε θα κινηθούμε. Ωστόσο, να σας πω ότι εμείς θεωρούμε ότι επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να επηρεάσουμε τα πράγματα στο Μαρόκο. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να εμβαθύνουμε περισσότερο συνεργασία με το Μαρόκο και να επανέλθουμε στην πρώτερη συνεργασία που είχαμε. Και θεωρούμε ότι η μετανάστευση είναι ένας μόνο από τους τομείς και νομίζω ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό και στον τομέα αυτό και στους υπόλοιπους τομείς να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία που είχαμε στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ πέρα, που μας ενημερώσατε.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 Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, α περάσουμε στο επόμενο σημείο τη σα διάταξη. Έχουμε μαζί μα ε, τον Επίτροπο για την Επιστημική Καινοτοπία και την Έρευνα, ο οποίος θα συζητήσει μαζί μας το ζήτημα της Science Diplomas, μονική διπλωματία και γιατί θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Γιατί θεωρώ ότι το έβρος της ε, διπλωματίας μας ε, θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι αυτό της κλασικής εξωτερικής πολιτικής. Και έτσι λοιπόν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθεί τα ε, συμφέροντά της και να προωθεί συγκεκριμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους ε, μέσω ακριβώς ε, ε, αυξημένης σύνδεσης και διπλωματικών ακριβώς σχέσεων και επιχειρηματικών σχέσεων. Γνωρίζουμε πως οι Αμερικανοί είναι πολύ επιτυχημένοι σε αυτό το επίπεδο, ότι έχουν επιτύχει μεγάλη πρόοδο και γνωρίζουμε ότι διάφορες πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιτύχει μεγάλες δραστηριότητες. Εδώ μεγάλες δράσεις και κάποιες είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και υπάρχει και ένα ακόμα σχετικό ζήτημα που είναι βέβαια διαφορετικό θεματικά, είναι το culture diplomacy, δηλαδή η ε, διπλωματία στο επίπεδο του πολιτισμού. Ένα τέτοιο είδος διπλωματίας μπορεί και αυτό πραγματικά να έχει ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο και ένα αντίκτυπο ο οποίο δεν περιορίζεται απλά και μόνο σε αυτή καθ' αυτή τη διπλωματία και ε, είναι λοιπόν και αυτό το είδο διπλωματίας πολύ ενδιαφέρον. Να δώσω όμως το λόγο στον Επίτροπο και τον ευχαριστώ που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ που με προσκαλέσατε. Είμαι ένας από τους πρώτους επιτρόπους για την επιστήμη, έρευνα και καινοτομία που έρχομαι εδώ στην επιτροπή σας αυτή. Και θέλω να σας πω ότι ειλικρινά σας ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως για την πρόσκλησή σας αυτή. Και αυτό γιατί όταν αρχίσαμε είχαμε την εντύπωση, μάλλον σκεφτόμαστε ποιοι είναι οι στόχοι της επιστήμης και της καινοτομίας αυτή τη δεκαετία. Και καταλήξαμε το ότι έχουμε τρία θέματα κυρίως. Πρώτον, άνοιγμα της καινοτομία, των επιστημών και άνοιγμα στον κόσμο. Άνοιγμα στον κόσμο είναι ακριβώ αυτός ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνα της στρατηγικέ μας στην καινοτομία και την έρευνα. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας μιλήσω ακριβώς για τις ιδέες αυτές που αναπτύσσουμε τώρα όσον αφορά τον πυλόν αυτό που τον ονομάζω εγώ άνοιγμα στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν στην Ευρώπη έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και ειδικό σκηνικό πικελομορφίας πρώτα απ' όλα που μας βάζει ε, πρώτους πρώτους στον κόσμο γιατί ακριβώ έχουμε τα συστατικά για να είμαστε πρώτοι. Να είμαστε πρώτοι στη θεμελιώδη έρευνα και στη συνέχεια την έρευνα αυτή την κάνουμε καινοτομία. Όταν λοιπόν η επιστημονική διπλωματία δεν είναι κάτι καινούριο στην Ευρώπη, παρόλα αυτά η έννοια παραμένει ακέραια. Και ένα από τα ζητήματα ε, τα οποία ε, χειρίζεται η Royal Society, μια που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την έννοια αυτή της επιστημονικής διπλωματίας, λέει λοιπόν η Royal Society ότι πρόκειται για μια ρευστή έννοια ακόμα. Τώρα θα σας πω ποιες είναι οι δικές μου απόψεις για την επιστημονική διπλωματία και πώς βλέπω εγώ όλα αυτά τα θέματα. Για μένα λοιπόν είναι ξεκάθαρα τα εξής. Πρώτον, ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις λύνονται μόνο με παγκόσμιες λύσεις. Και δεύτερον, σήμερα καμία χώρα από μόνη της, κανένας επιστήμονας, κανένας άνθρωπος, καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι αν κοιτάξετε το 1911 όταν είχαμε το πρώτο τεκμήριο για την ιδέα, τη θεωρία αυτή των κυμάτων βαρύτητας, αυτό το επιστημονικό έγγραφο είχε ένα συντάκτη μόνο, τον Einstein. Σήμερα όμως το 2016 αυτό το οποίο αποδεικνύει το σωστό της θεωρίας εκείνης υπογράφεται από πάνω από χίλιους διαφορετικούς συντάκτες και από πάρα πολλές χώρες. Αυτό ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά πώς η επιστήμη προθεί το πριν από χίλια χρόνια και πως σήμερα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα αυτές τις προκλήσεις της επιστημονικής ε, διπλωματίας. Μπορούμε να τα δούμε αυτά τα ζητήματα από τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η πρώτη είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες και να βελτιώσουμε τις διεθνείς σχέσεις. Η Royal Society πάλι το ονομάζει αυτό επιστήμη στην υπηρεσία της διπλωματίας. Το δεύτερο είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, τις οποίες αναφέρθηκα πριν, μέσω της επιστημονικής συμβουλής, δηλαδή επιστήμη στη διπλωματία. Και το τρίτο είναι βέβαια η υποστήριξη της παγκοσμιοποίησης μέσω παγκόσμια συνεργασία στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία. Θα σα πω τώρα ποια είναι τα σχέδιά μα και τι κάνουμε για το πρώτο, δηλαδή για αυτό το γεφύρωμα για να βελτιωθούν οι διεθνείς σχέσεις. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έπρεπε να κάνω ήταν να υπογράψω μια συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία ε, και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμά μας Horizon 2020. Και ήταν μια μοναδική στιγμή έβλεπε όλους αυτούς τους επιστήμονες και τους ερευνητές της Ουκρανίας, τόσο ταλαντούχους, οι οποίοι διψούσαν για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμά μας, οι οποίοι μας το ζητούσε και μας λέγαν πόσο καλά πράγματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, κάτι το οποίο δεν ακούμε τόσο συχνά στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη λέμε το 2020 το Horizon είναι πολύ μεγάλο σημαντικό πρόγραμμα κτλ. Αλλά αν πάτε σε μια χώρα σαν την Ουκρανία, τότε είναι που νιώθετε ότι είναι πραγματικά σημαντικό. Και για αυτούς, περισσότερο και από τα χρήματα τα οποία παίρνουν, ε, σημασία έχει το δίκτυο. Και μετά προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο και συμπεριλάβαμε και την Τινησία. Και αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί με την υπογραφή αυτή της συμφωνίας ε, ρίξαμε γέφυρες και σε μια χώρα η οποία και αυτή με φοβερό ενθουσιασμό θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμά μας. Πέρα από αυτές τις δύο συμφωνίες που ήταν δύο πολύ σημαντικές στιγμές πέρυσι, η πιο σημαντική γέφυρα που δημιουργήσαμε και για την οποία είμαι πολύ περήφανος ήταν ότι πήγαμε στον πρώτο επιταχυντή σωματεδίων της Μέσης Ανατολής. Έχουμε στην Ευρώπη έναν, αλλά και στο Μαν, στην Ιορδανία υπάρχει ένας άλλος. Και όταν πήγα εκεί, ένιωσα ότι ζούσα μια μαγική στιγμή. Ήμουνα σε αυτή τη συνάντηση με επιστήμονες από το Ισραήλ που καθόντουσαν δίπλα-δίπλα με επιστήμονες από την Παλαιστίνη και άλλους από το Ιράν, επιστήμονες οι οποίοι συνεργαζόντουσαν με έναν νέο από το Πακιστάν, ο οποίος ήταν εκεί για το PhD του το διδακτορικό του. Εμείς ήμασταν παρατηρητές λοιπόν εκεί και συνεισφέρουμε και πρέπει να πω ότι είμαστε το θεμελιώδες στοιχείο του προγράμματος αυτού. Σε λίγο θα πω και στο Ιράν. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο διαλόγου, επιστημονικού διαλόγου μαζί τους και να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα μέσα για το διάλογο αυτό. Και τέλος όσον αφορά τις γέφυρες αυτές που χτίζουμε, υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που είναι μέρος του μέλλοντός μας στην ε, Μεσόγειο και αυτό είναι το πρίμα. Είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που φτιάξαμε με μεσογειακές χώρες όσον αφορά ε, τα τρόφιμα και το νερό. Πώς λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε με όλες τις μεσογειακές χώρες και να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερη έρευνα στον τομέα των τροφίμων και να το συνδέσουμε με τον ψηφιακό κόσμο. Για μένα Όλα αυτά είναι οι γέφυρες οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα στο μέλλον γιατί θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις προκειμένου να περάσουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας τώρα βασίζεται στο εξή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις μέσω σωστών ε, επιστημονικών ε, συμβουλών. Εμείς το πρώτο χρόνο αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο τέτοιων επιστημονικών ε, συνεργασιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό που ονομάσαμε Επιστημονικό Συμβουλευτικό Μηχανισμό. Εφτά από τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο δίνουν το χρόνο τους για να συνεργάζονται μαζί μας και βοηθούν τους πολιτικούς στις αποφάσεις τους σε διάφορα ζητήματα. Αν λοιπόν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αν η Κομισιόν πρέπει να πάρει μια απόφαση, πρέπει να έχουμε στοιχεία από τον επιστημονικό κόσμο και βάσει αυτών να αποφασίζουμε. Εφτά λοιπόν από τους καλύτερους επιστήμονες έχουμε εμείς. Ένας είναι ένας που ήταν γενικός διευθυντής της ΕΡΝΑ. Έχουμε έναν λαμπρό Γάλλο μαθηματικό και εδώ κοιτάω προς την Υπουργό Λιωμαρή, τι θυμάμαι, και πολλούς άλλους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας προσφέρουν το χρόνο τους για να μας βοηθήσουν ε, με επιστημονικά δεδομένα να πάρουμε τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε σε δύσκολες αποφάσεις στο μέλλον. Τον πρώτο χρόνο είχαμε δύσκολες καταστάσεις. Είχαμε την επιθυμία έμπολα που ξέσπασε στη Δυτική Αφρική και ε, μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να αντιδράσει γρήγορα με αυτή την κρίση, ενώ έπρεπε να αντιδράσουμε γρήγορα. Τελικά, σε δύο μήνες μπορέσαμε, συνδέοντας δημόσιους πόρους και ιδιωτικούς ε, πόρους, να βρούμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ και κανένας δεν ήξερε τι έγινε με αυτά τα χρήματα. Όμως ένα από τα εμβόλια τα οποία δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπιστεί ο ιός έμπολα ε, το εμβόλιο αυτό δημιουργήθηκε με τα χρήματα αυτά των ε, Ευρωπαίων φορολογούμενων και του ιδιωτικού τομέα. Και έτσι έχουμε περάσει τώρα στις κλινικές εφαρμογές ε, στα 2-2. Έχουμε λοιπόν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη, που δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν τα γενοποιούμε αρκετά, δεν γίνονται γνωστά στον κόσμο. Και όμως, ήμασταν ένα σημαντικό κομμάτι της λύσης για την επιδημία έμπολα. Επίσης ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το διακυβερνητικό πάνελ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, το IPCC. Και εκεί εμείς, η Γενική Διεύθυνση για την Έρευνα και την Καινοτομία, έχει τα στοιχεία τα οποία πηγαίνουν σε αυτό το πάνελ. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να βοηθήσουμε τους πολιτικούς μας όταν διαπραγματευόμαστε, ώστε να ξέρουν ποια είναι τα στοιχεία τα ακριβή στοιχεία που χρειάζεται το IPCC και πολλά από αυτά προέρχονται από εμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα υπάρχει και η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση. Εδώ αναπτύξαμε και ένα πρόγραμμα που λέγεται Επιστήμη για τους πρόσφυγες και θέλω να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό. Θελήσαμε δηλαδή να αντιστοιχίσουμε τους θεσμούς που θέλουν να βοηθήσουν με τους μετανάστες που είναι ερευνητές και επιστήμονες και που έχουν ανάγκες. Εκατό τέτοια ιδρύματα επιστημονικά είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν. Σήμερα έχουμε 224 ερευνητικές οργανώσεις που έχουν πει ότι έχουν θέσεις για μετανάστες και έχουμε 42 ερευνητές πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ε, δηλωθεί στην ιστοσελίδα αυτή. Εμείς συνεισφέραμε προκειμένου να βρεθεί αυτή η σύνδεση ε, μεταξύ των ανθρώπων και οι άνθρωποι αυτοί που είναι ταλαντούχοι αλλά βρίσκονται σε μια απελπιστική κατάσταση ανθρωπιστικά να μπορέσουν να βοηθηθούν ως ερευνητές. Έρχομαι στο τρίτο σκέλος τώρα της στρατηγικής μας που είναι πραγματικά η διπλωματία για την επιστήμη. Η έρευνα και η καινοτομία γίνεται και εκτός Ευρώπης βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις δικές της γνώσεις και βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα, δεδομένου ότι εμείς διαθέτουμε γνώση επιστημονική και ερευνητική και είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στον κόσμο. Και πριν από το 7ο ε, πρόγραμμα έρευνας είχαμε 170 χώρες που συμμετείχαν με 5.167 συμμετέχοντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως τώρα προσπαθεί να βρει πού βρίσκεται το ταλέντο και να συνεργαστεί. Ένα βασικό θέμα για την επιστήμη σήμερα είναι ότι δεν αφορά έναν άνθρωπο, δεν είναι ατομικό. Δεν έχει να κάνει ούτε με μία επιστήμη, έχει να κάνει με συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών τομέων. Υπογράψαμε λοιπόν με την Κίνα έναν μηχανισμό χρηματοδότηση, 30 εκατομμύρια βάζει Κίνα κάθε χρόνο και εμεί με το Ράζο 2020 συνεισφέρουμε για να έχουμε περισσότερους Κινέζους επιστήμονες εδώ και περισσότερους Ευρωπαίους επιστήμονες στην Κίνα και με το Μεξικό και με την Νοτιά Κορέα, με την Ιαπωνία, με κάποιες περιοχές στη Βραζιλία. Συνεργαζόμαστε και το 2014 η συνεισφορά φτάνει στα 16 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να στηρίξουμε αυτήν την παγκόσμια διάσταση της διπλωματίας για την επιστήμη. Ξέρετε ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ τελευταία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Τώρα πρέπει να περάσουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο που να είναι η παγκόσμια έρευνα με συγχρηματοδότηση, με μηχανισμούς, αποφάσεις που έχουμε πάρει δηλαδή ήδη από τον Ιούνιο του 2015 έχουμε καταφέρει να μπούμε με τις χώρες ΣΕΛΑΚ σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πλαίσιο συνεργασίας στην έρευνα. Βλέπετε ότι η Ανατολή και προσπαθούν να προχωρήσουν, να βοηθήσουν τους επιστήμονες να μετακινούνται ανά τον κόσμο. Αυτό είναι ζωτική σημασία για να έχουμε καλύτερη επιστήμη. Πολλές φορές λοιπόν με ρωτάει ο κόσμος και μου λέει «Μα δεν φοβάσαι ότι τελικά δίνεις γνώση σε άλλους» Ναι, αλλά εγώ απαντάω ότι αν δεν μοιραστεί τι γνώσει σου με του υπόλοιπου, δεν έχει επιστήμη. Άρα χρειάζονται τα δίκτυα αυτά, όπου και οι άλλοι θα σου δίνουν εσένα πληροφορίε και γνώση, αλλά και εσύ θα δίνει γνώση στους άλλους. Ανταλλάσσουμε ιδέες. Κάποιες ιδέες που μπορεί να είναι δικές σου, μπορεί να πρέπει να τις προστατεύσεις, αλλά τη γνώση πρέπει να την ε, μοιράζεσαι με τους άλλους. Εξάλλου, ε, μην ξεχνάτε ότι η σύμβαση ΣΕΡΝ επικυρώθηκε το 1954, τρία χρόνια πριν από τη συνθήκη της Ρώμης. Και σήμερα λοιπόν θα κλείσω με τα λόγια του Σερ Τζόζεφ Μπάνξ, Βρετανός φυσιοδήφης, ο οποίος ε, παρέμεινε σε επαφή με τον Μπέντζαμιν Φράγκλεν, ακόμα και όταν ο Φράγκλεν είχε υπογράψει τη δήλωση ανεξαρτησίας και έγινε εκτρός του Ηνωμένου Βασιλείου. Και είπε ότι η επιστήμη δύο εθνών μπορεί να είναι σε καλές σχέσεις παρόλο που οι πολιτικοί μπορεί να βρίσκονται σε πόλεμο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που μου δώσετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την επιστημονική διπλωματία. Τους μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ε, κύριε Σας, ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τα όσα μας είπε μόλις τώρα ο Πέτροπος, τον ευχαριστώ για το γεγονό ότι έχει αναγνωρίσει πράγματι τη μεγάλη σημασία της ε, επιστημονικής ε, διπλωματίας. Υπάρχει ε, βέβαια κάποια αντίσταση ό,τι αφορά τη διεύρυνση αυτού του ορισμού, αν θέλετε, της δημοκρατίας, για παράδειγμα και με την πολιτισμική διπλωματία. Όμως η διπλωματία της σήμερα ημέρα θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με άλλες πολιτικές, δηλαδή και η πολιτισμική διπλωματία θα πρέπει να συνδεθεί και με την επιστημονική διπλωματία γιατί η σύγχρονη ε, διπλωματία ε, αντί να ε, συμβάλλει στο να έρθουν οι λαοί πιο κοντά μεταξύ τους, πολλές συχνές έχει συμβάλλει στο να οξύνει τις καταστάσεις να, να, γίνουν ε, να, στην, στις σειράξεις και διάφορα είδη πολέμων έχουν υποστηριχθεί αν θέλετε η δημοκρατία. Άρα λοιπόν θα πρέπει με την επιστημονική διπλωματία όπως είδαμε και με την ίδια την επιστημονική έρευνα να, δημιουργούνται, να δημιουργείται τέτοια δικτύωση και να δημιουργείται και μια διεθνής επιστημονική κοινότητα. Και έτσι λοιπόν το πώς μπορεί να μας υπηρετήσει αυτή αυτή η επιστημονική κοινότητα μέσα τη επιστημονική διπλωματία είναι πολύ σημαντικό. Ειδικότερα αυτό αφορά περιοχέ ε, του κόσμου τι οποίε έχουμε δύσκολη πρόσβαση. Έτσι λοιπόν η επιστημονική διπλωματία εδώ μπορεί να μα βοηθήσει να ε, επιτύχουμε κάποια πρόοδο γιατί είμαστε πιο ανεπτυγμένοι στο επίπεδο τη επιστημονική έρευνα. Και εδώ αναφέρομαι για παράδειγμα στη συνεργασία με χώρε τη Λατινική Αμερική. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για συνεργασία αλλά και με άλλε περιοχέ του κόσμου μπορούν να γίνουν περισσότερα. Ένα τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω στον Επίτροπο. Ε, ε ποια είναι η στάση που έχετε αντιμετωπίσει, αν θέλετε, από πλευρά του Συμβουλίου, από τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά ακριβώ την προώθηση αυτή τη επιστημονική διπλωματία. Είναι διατεθειμένα πράγματι να δώσουν περισσότερη αξία σε αυτή την επιστημονική διπλωματία. Σα ευχαριστώ πολύ. Euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο γιατί η παρουσίασή του ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκεκριμένη και παρουσίασε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Ένα ερώτημα όμως, όταν, μιλήσετε, όταν μιλήσατε για την υφιστάμενη, τη μελλοντική συνεργασία, αναφερθήκατε στην Κίνα, στη Μέση Ανατολή, αναφερθήκατε σε ορισμένες χώρους ουσιαστικά οι οποίες υστερούν μπορούμε να πούμε κάπως ε, στην έρευνα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναφερθήκατε καθόλου σε ενδεχόμενη συνεργασία επιστημονική με τη Ρωσία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με χώρες δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την επιστημονική έρευνα. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν τι προβλέπετε να κάνετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες αυτές, προκειμένου η επιστημονική μας συνεργασία να είναι κάπως πιο ισορροπημένη. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι η συνεργασία που έχουμε μάλλον είναι ανισόρροπη και δει εις βάρος μας. Κύριε Γκάμπριελ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, για τις ιδέες που εκφράσατε. Δύο ερωτήματα θέλω να θέσω. Πρώτον, σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Αλιό Μαρή, θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στην Μεσόγειο. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα Εράσμους ειδικά για την περιοχή της Μεσογείου. Νομίζω ότι το ζήτημα που τίθεται εμπροκειμένο δεν είναι ζήτημα χρηματοδότησης, αλλά πολιτικής σημασίας. Και ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι στην περιοχή αυτή του κόσμου που περιμένουν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεύτερον, είπατε ότι η ευρωπαϊκή διπλωματία θα πρέπει να λάβει υπόψη της την επιστημονική διπλωματία. Η επιστημονική όμως κοινότητα δείχνει την ανάλογη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ποια πλατφόρμα θα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να συνεργαστείτε με τους ε, ευρωπαίους επιστήμονες και ερευνητές και προκειμένου πραγματικά βασιζόμενοι στην επιστήμη να καταφέρετε να προασπίσετε τα πολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω καταρχάς πορτογαλικά και στη συνέχεια γαλλικά, απαντώντας σε ερωτήσεις αυτές. Απευθυνόμενο στον ε, κύριο Φρανσίσκο Ασής, ε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για τα λόγια σας ε, και για την υπενθύμηση που μας κάνετε σε ό,τι αφορά το ρόλο της επιστήμης και τα όσα σχολιάσετε περαιτέρω σε ό,τι αφορά τη σημασία, τη σημασία της. Πράγματι, ε, θα ήθελα να βασιστώ στα λόγια που είπε ο κύριο Ασίσο δηλαδή είμαστε πραγματικά εξαιρετικά ανεπτυγμένοι στο πεδίο τη έρευνα. Ε, ε, δηλαδή, δεν γνωρίζουμε συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 7 εκατομμύρια επιστήμονε παγκοσμίω, το 22% εντοπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράγουν αυτή, αυτό το 22%, το 30% της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης και ε, το 1 τρίτο των ε, παραπομπών που γίνονται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις αφορούν ε, δημοσίευσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης μου έδωσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, δηλαδή με ποιο βαθμό έχει γίνει δεκτή αυτή η πρωτοβουλία για την επιστημονική διπλωματία από το Συμβουλίο και τα κράτη-μέλη. Νομίζω πως έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως προς την ευθυγράμμιση της τάσης των διαφόρων κρατών μελών σε σχέση με αυτήν την περαιτέρω ανάπτυξη και την επικοινωνία στο επιστημονικό επίπεδο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ένα ε, μέσο άσκησης της διπλωματίας. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών ε, σήμερα και νομίζω πως οι υπουργοί ε, για τις επιστήμες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν περισσότερο σε αυτό το επίπεδο και να συμπεριλαμβάνονται σχετικές συζητήσεις για τη διπλωματία. Για παράδειγμα, εγώ θέλω πάντοτε ή είπατε εκπρόσωπο ε, για τα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική ε, ε, τη Επιτροπή, κυρία Μοντιρέ, να με προσκαλεί πάντοτε στι συνεδριάσει τη ω εγώ επίτροπο τη έρευνα. Και αυτό νομίζω αυτή η, η στάση θα πρέπει να υιοθετηθεί και από όλου του υπουργού για ε, ε, ζητήματα επιστημών στα διάφορα ε, κράτη-μέλη απέναντι στου υπουργού εξωτερικών. Απαντήσω τώρα στην κυρία Μισελ Αλιομαρίου όσον αφορά το ζήτημα τη συνεργασία. Το ερώτημά σας είχε να κάνει με συνεργασία που θα μπορούσαμε να είχαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες περιοχές του κόσμου. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια πάρα πολύ καλή και έντονη συνεργασία σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας. Έχουμε μάλιστα ένα πρόγραμμα συνεργασίας ιδιαίτερα εμβαθυμένο με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, National Institute of Health των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επίσης και με άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ισότιμη η συνεργασία που έχουμε. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που διαβλέπω εγώ. Στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, όντως ε, έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα και είναι ακριβώς αυτός ο ψηφιακός τομέας που θα πρέπει να περάσει πλέον στην κλασική συνηθισμένη βιομηχανία. Τον κλάδο δηλαδή τη βιομηχανία που εκπροσωπούμε εμεί πάρα πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πέρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Για παράδειγμα στις νέε μορφέ βιομηχανία, στον κλάδο βιομηχανία 4.0 ή στον τομέα της φυσικής για παράδειγμα. Ακριβώς λοιπόν επειδή εμείς είμαστε ιδιαίτερα αναπτυγμένοι όσον αφορά την βιομηχανία, την κλασική βιομηχανία, μπορούμε να αποφεληθούμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά το ψηφιακό τομέα, προκειμένου να καταστήσουμε τη δική μας βιομηχανία πιο ψηφιοποιημένη. Και βλέπω επίσης, εξετάζοντας διάφορα αριθμητικά δεδομένα, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό του προπολογισμού μας έχει να κάνει με τις επενδύσεις στον τομέα αυτό, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε από την άλλη έχουν κάνει πολύ σημαντικότερες επενδύσεις στο ψηφιακό τομέα. Τώρα, όσον αφορά τη Ρωσία, Επί του παρόντος προσπαθώ να δω αν θα μπορούσα σύντομα να πάω στην Ρωσία προκειμένου μέσω περαιτέρω επαφών να συνεχίσουμε την ιστορική επιστημονική συνεργασία που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας αν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα που είχαμε πριν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, υπάρχει σαφώς μία μείωση στην, στον αριθμό των επαφών αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εντείνουμε και να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους Ρώσους επιστήμονες. Ετέθη ένα ακόμα ερώτημα από την κυρία Γκάμπριελ, η οποία αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Εράσμους. Όπως το γνωρίζετε, εγώ είμαι γέννημα θρέμα του προγράμματος Εράσμους. Προφανώς είμαι ενθουσιώδης υπερασπιστής του προγράμματος αυτού και θα διαβιβάσω το μήνυμά σας στον Επίτροπο Τίμπορ Ναβάσκιτς, ο οποίος είναι αρμόδιος για ζητήματα πολιτισμού και παιδείας. Νομίζω ότι όντως το σχέδιο αυτό στο οποίο αναφερθήκατε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους νέους. Και εγώ θα κάνω κάθε το δυνατό προκειμένου να καταφέρω να συμβάλλω από τη δική μου τη θέση για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Θα διαβιβάσω πάντως στον ε, συνάδελφό μου το μήνυμά σας. Και θέσατε ένα ακόμα ερώτημα που έχει να κάνει με τους ε, επιστήμονες ε, το πόσο μπορούν να βαρύνουν στις πολιτικές αποφάσεις. Ξέρετε, πολύ συχνά οι επιστήμονες ε, δεν καταφέρνουν να επικοινωνήσουν πάρα πολύ καλά. Μιλάω πολύ συχνά με επιστήμονες και τους λέω ότι αν καταφέρνατε να προβάλλετε με έναν τρόπο εκλαϊκευμένο το έργο σας, τότε πραγματικά θα μπορούσε να επηρεάσετε πάρα πολύ την πορεία που ακολουθεί ο κόσμος αυτός. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολλοί ερευνητές, πολλοί επιστήμονες που συντοποιούν αυτή τους τη δύναμη και αρχίσουν και εντάσσουν περισσότερες προτεραιότητές τους την ε, καινοτομία. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλέ κυβερνήσει οι οποίε δεν είχαν συνειδητοποιήσει στο παρελθόν τη δύναμη τη επιστήμης και τη καινοτομία. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί που αρχίζουν και συνειδητοποιούν πόσο πολύ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα με τη χρησιμοποίηση τη επιστήμης και τη καινοτομία. Ακριβώ αυτό κάνουν και οι Κινέζοι. Πρόσφατα, ακούγοντα ε, τον Πρωθυπουργό της Κίνας ε, συνειδητοποίησα ότι ένα μεγάλο μέρος του λόγου του αναφερόταν ακριβώς στην επιστήμη και στην καινοτομία. Νομίζω ότι χωρίς καινοτομία και χωρίς επιστήμη και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε ποιοτικά να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έδωσε σήμερα εδώ. Ε, νομίζω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε την ασχόλησή μας με αυτό το ζήτημα τόσο σε ό,τι αφορά δηλαδή την επιστημονική διπλωματία αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική στο επίπεδο του πολιτισμού και την πολιτισμική διπλωματία. Ίσως θα μπορούσαμε κατά την επόμενη συνέντευξη του Προεδρείου να εξετάσουμε το πώς ε, μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτή την ε, ανεργοποίησή μας σε αυτό το επίπεδο και καλό θα ήταν να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά τον Επίτροπο που βρήκε το χρόνο να έρθει σήμερα εδώ και εύχομαι σε όλους καλό μεσημέρι.